Well, Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε. Έχετε λάβει την ημέρη σε διάταξη. Έχετε μήπως παρατηρήσει να μπορούμε να την εγκρίνουμε. Όπως ξέρετε, σήμερα συνεδριάζει το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών με θέμα την Ουκρανία μετά το δημοψήφισμα στην Κρυμαία. Έχουμε ήδη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών και το βασικό θέμα είναι ότι ελήψη αποτελεσμάτων, γιατί έγινε μια προσφορά όπως ξέρετε, ελήψη αποτελεσμάτων, το Συμβούλιο αποφάσισε να θεσπίσει επιπρόσθετα μέτρα καθώς και περιορισμό μετακινήσεων και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για για ανθρώπους που, ε, για τους οποίους υπάρχουν υπόνοιες ότι υπονομεύουν την κυριαρχία και την ενταφική αικαιρότητα της Ουκρανίας. Θα σας ε, μοιράσουμε τα συμπεράσματα αυτά και ίσως αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε πιο διεξοδικά. Μπορεί να προσκαλέσουμε και τον κύριο Βημό για την αυριανή συνεδρίαση. Πρακτικά πρακτικά της συνεδρίασης της 21ης ε, Ιανουαρίου υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι, οπότε εγκρίνονται. Περνάμε στο πρώτο σημείο της ημερήσης διάταξης, τη δημόσια ακρόαση σχετικά με την απάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εξωτερική και εμπορική πολιτική της Ρωσίας έναντι των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ τον κύριο Βαγουένσα, τον συνάδελφο που εκπροσωπεί εδώ την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και θα παρακολουθήσει την δημόσια κρόση. Θα συζητήσουμε κάτι, ένα θέμα δηλαδή που πριν τις εξελίξεις στην Κρυμαία ήδη ήταν αρκετά ανησυχητικό. Και εννοώ τα μέτρα που έλαβε η Ρωσία κυρίως τα εμπορικά και των οικονομικών σχέσεων ε, ε, στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Θα πρέπει να λάβουμε θέση για τα θέματα αυτά υπό το φως των νέων των χθεσινών εξελίξεων μετά την έκβαση του δημοψηφίσματος στην Κρυμαία και την ε, ανάγκη να αντιδράσουμε κάπως σε όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν τέσσερις εμπειρογνώμονες, την κυρία, τη δόκτωρα Βόλτσουκ, που ε, έρχεται από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ. τον κύριο Καζιέ, από τη Σχολή των Βρυξελών για τις Διεθνείς Σπουδές και το Πανεπιστήμιο Κέν των Βρυξελών. Έχουμε τον κύριο Βίγκαντ, που είναι διευθυντή στην Υπηρεσία Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και τον κύριο Μπάλα από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Βαγουένσα τον εκπρόσωπο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου εδώ στην Δημόσια Κρόση. Σας ευχαριστώ, χαίρομαι για αυτή την ε, ε, συνδιοργάνωση που γίνεται από τις δύο επιτροπές της δημόσιας ε, αυτής ακρόση, που είναι πολύ επίκαιρη δυνάμει και των εξέλιξεων. Σε ό,τι αφορά την ανατολική εταιρική σχέση που ξεκίνησε το 2008, οι Ευρωπαίοι θεωρούν την, εταιρική αυτή, την ανατολική εταιρική σχέση ως κινητήριο μοχλό για μεταρρυθμίσεις στι έξι αυτές χώρες τη εταιρική σχέσης. Ενώ έχει αντιμετωπιστεί ω απειλή αυτή η εταιρική σχέση από τη Ρωσία ή θεώρησε την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ως αντίπαλο στα δικά της σχέδια όπως είναι η Ευρασιακή Τελωνιακή Ένωση. Η Ρωσία λοιπόν φυσικά δεν θα ήταν ε, μέλος αυτής της εταιρική σχέσης. Επιπλέον όμως δεν θα άφηνε και τους στενότερους εταίρους όπως την ε, Λευκορωσία να λάβουν μέρος σε αυτή την ανατολική εταιρική σχέση. Και όσο μεγάλωναν οι φιλοδοξίες αυτής της εταιρική σχέσης, και φτάσαμε προς την τελική της φάση, τους τελευταίους μήνες ε, γίναμε μάρτυρες μιας εντατικοποίησης των μέτρων της Ρωσίας που είχαν στόχο να πείσουν τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης να εγκαταλείψουν την εταιρική αυτή σχέση και τη συμφωνία σύνδεση, ε, χάρη μια φιλορωσικής πολιτική ε, και τη προσχώρησή του στην Ευρασιατική Τελωνιακή Ένωση. Αυτό ξεκίνησε με, αδικαιολόγητες, ε, με αδικαιολόγητους εμπορικούς περιορισμούς απέναντι στην Ουκρανία και τη Μολδοβία πέρυσι το καλοκαίρι. Συνεχίστηκε με πολιτικές πιέσεις στην Αρμενία και τη Γεωργία με βάση τις δικές τους ανησυχίες ε, για την ασφάλεια και με χρηματικ... Ε, δημοσιονομικές και χρηματοοικονομικές πιέσεις προς την Ουκρανία. Μετά την αλλαγή της Ουκρανικής κυβέρνησης ε, είχαμε ακόμη μεγαλύτερες εξελίξεις, ιδίως πιθανή προσάρτηση της Κρυμαίας στη Ρωσία, κάτι που διακυβεύει όχι μόνο τις ρωσο-ουκρανικές σχέσεις, αλλά και το την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις διεθνείς διπλωματικές σχέσεις. Βέβαια σε κάποιο βαθμό όλοι περιμέναμε ότι η Ρωσία δεν θα άφηνε να στεφτεί με επιτυχία η Σύνοδος Κορυφής του Βίλνιους ή δεν θα άφηνε τους διαδηλωτές του Μαϊντάν να πετύχουν μια ειρηνική δημοκρατική μετάβαση στην Ουκρανία. Η Ρωσία λοιπόν ήθελε να εκτροχιαστεί η ανατολική εταιρική σχέση χρησιμοποιώντας την εξουσία της σε διάφορα επίπεδα, στις τιμές ενέργειας, ασκώντας πιέση εμπορικά θέματα, ασκώντας πολιτικές πιέσεις στις συμμάχους στις ε, γειτονικέ χώρες, δημιουργώντας κάποιες ε, εντάσεις στο τομέα της ασφάλειας και ούτω καθεξής. Οι ρωσικές πολιτικές μέχρι στιγμής ε, ε, είχαν κάποια επιτυχία και δημιούργησαν προβλήματα που κατά τη γνώμη και θέματα που κατά τη γνώμη θα πρέπει να τα αναλύσουμε σήμερα. Γιατί λοιπόν αυτές οι χώρες υπέκυψαν στις ρωσικές πιέσεις. Θα πρέπει να αντιληφθούμε την δέσμευσή τους προς την ε, ε, ανατολική εταιρική σχέση να έχει εξασθενήσει Κάτι που δείχνει διαρθρωτικές αδυναμίες σε οικονομικά θέματα και θέματα ασφάλειας. Αδυναμίες δηλαδή της ανατολικής εταιρικής ε, σχέσης. Πώς λοιπόν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί καλύτερα, να αντιδράσει καλύτερα στις ρωσικές πολιτικές που στόχο έχουν την παρεμπόδιση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες. Έχουμε κάποιους μηχανισμούς και εργαλεία για να βοηθήσουμε τις χώρες ανατολικής εταιρικής σχέσης. Αυτού τους μηχανισμούς και αυτά τα εργαλεία θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε πιο συχνά, να τα βελτιώσουμε ή και μερικές φορές να τα μεταρρυθμίσουμε άρδιν. Επίσης μπορούμε και επικοινωνιακή εκστρατεία να έχουμε για να εξοδετερώσουμε την αντίστοιχη επικοινωνιακή προσπάθεια της Ρωσίας στις χώρες Ανατολικής Γειτονίας και Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Έχουμε λάβει αρκετά μαθήματα τους τελευταίους μήνες γιατί και εκεί έχουμε πολλές αδυναμίες. Τέλος, στο παρόν πλαίσιο της εισβολής της και παρέμβασης της Ρωσίας στην Κρυμαία, διαρωτόμαστε αν ήταν επαρκή η αντίδραση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα το πακέτο συνδρομή που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που το ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προ την Ουκρανία είναι ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση για να επανέλθει η Ουκρανία στο δρόμο της οικονομικής ανάκαμψης, αλλά είναι επαρκές ένα τέτοιο μέσο για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος στην ασφάλεια. Θα υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία. Ακόμη και αν το κάνει όμως, ε, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα επανέλθει η Κρυμαία στην, Ουρανι... στην Ουκρανική κυριαρχία. Είναι όλα αυτά σημαντικά ερωτηματικά και απορίες που θα κληθούμε να απαντήσουμε σήμερα και ελπίζω ότι οι καλεσμένοι μας, ε, που είναι και πανεπιστημιακοί σε πολλές περιπτώσεις, θα μας δώσουν κάποιες ενδείξεις και κάποιες ε, απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα, ώστε να αποτρέψουμε την επανάληψη τέτοιων πιέσεων στο μέλλον. Και αν μου επιτρέπετε, θα Κάνω εγώ την εισαγωγή και θα σας παρουσιάσω τους καλεσμένους μας. Ευχαριστώ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στη δόκτωρα Βόλτσουκ και επειδή έχει παρουσίαση με PowerPoint θα την καλούσα στο βήμα. Παρακαλώ να περιοριστείτε σε ένα δεκάλεπτο στις παρεμβάσεις μας για να έχουμε χρόνο για συζήτηση. Η κυρία Βόλτσουκ, η δόκτωρ Βόλτσουκ έχει το λόγο. Um, Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, είναι επίκαιρη η σημερινή συζήτηση. Θα μιλήσω για τη Ρωσία και τις οικονομικές επιπτώσεις της πολιτικής της, πώς μπορεί να επηρεάσει τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας η Ρωσία και τι κίνητρα μπορεί να δώσει, πώς μπορεί να τιμωρήσει εφόσον ακολουθούν την ευρωπαϊκή πορεία, για να το πούμε έτσι. Είμαι πολιτική επιστήμων, οπότε θα, θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τους οικονομολόγους στην αίθουσα, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να έχει κανείς μια πολιτική άποψη για τα πράγματα ως επιστήμων, διότι η συμπεριφορά της Ρωσίας προς τους εταίρους μας της Ανατολικής Γειτονίας έχει να κάνει πάρα πολύ με την πολιτική και το κράτος δικαίου στη Ρωσία, το πώς συμπεριφέρεται δηλαδή η Ρωσία ως διεθνής πρωταγωνιστής. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια συμπεριφορά. Όμως ως πολιτική επιστήμον μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι η Ρωσία όχι μόνο απλώς θα ξεκινήσει, αλλά έχει ήδη αρχίσει να τιμωρεί τους εταίρους από οικονομικής πλευράς. Ωστόσο, με διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικούς στόχους. Και θα εξηγήσω τι μπορεί να γίνει από την πλευρά της Ρωσίας θα επικεντρωθώ στην Γεωργία, την Ουκρανία και την Μολδαβία. Και θα ξεκινήσω με το ευρύτερο πλαίσιο γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που ίσχυε στο 2010 στην, ε, μετά, στην περιοχή της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ήταν μια πολύ ευέλικτη, επιλεκτική ε, και χαλαρή σύνδεση οικονομικών σχέσεων. Υπήρχε μια σειρά από συμφωνίε διμερεί και κάποιοι το ονόμαζαν αυτό ένα πιάτο με σπαγκέτι. Υπήρχαν ε, μια σειρά από ε, συμφωνίε λοιπόν πολυμερεί και διμερεί στον πρώην Σοβιετικό χώρο. Επίση, υπήρχε μικρό βαθμός εκπροσώπηση και πολύ χαμηλή ε, επιβολή του νόμου και υλοποίηση. Οι χώρες αυτές αποφάσιζαν τις εμπορικές τους σχέσεις με πολύ ευέλικτο και διαλλακτικό τρόπο. Αυτό ήταν το ευρύτερο πλαίσιο. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Τελωνιακή Ένωση της Ευρασίας με τον ενιαίο οικονομικό χώρο που αναμενόταν για το 2015, αυτή η Ευρασιατική Τελωνιακή Ένωση έχει αλλάξει πολύ, διότι ε, προβλέπει ένα καθεστώς αυστηρότερων νόμων για βαθύτερη οικονομική ε, ένωση στον πρώην Σοβιετικό χώρο. Ε, εδώ θα αναφερθώ και στον, θα απευθυνθώ στον κύριο Βαλέσα, διότι είναι σημαντικό αυτό για την μετέπειτα συζήτησή μας. Πώς ε, αποκρίθηκε, ανταποκρίθηκε η Ρωσία στην ανατολική γειτονία αυτή καθεαυτή και στα πλαίσια της αναμενόμενης Ευρασιατικής Τελωνιακής Ένωσης. Γιατί τώρα έχει σημασία αυτή η Ευρασιατική ολοκλήρωση, τι καθεστώς ισχύει. Όπως έλεγα, είναι ένα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα επιχείρημα για βαθύτερη οικονομική ε, σύνδεση που χαρακτηρίζεται από διαφορές και αποκλίσεις μεταξύ των κρατών και από την πλευρά του οικονομικού τους δυναμικού αλλά και ως προς το πολιτικό σκηνικό ε, επιβάλλεται στο Καζακστάν και στη Βινή Λευκορωσία η Ρωσία ούτως ή αλλά και η κάθε χώρα θα έχει μία ψήφο σε αυτή τη μετέπειτα ένωση. Οπότε μπορεί να καταψηφιστεί κάτι που προτείνει η Ρωσία. Ε, λόγου χάρη για του δασμού. Οι δασμοί που επιβάλλει η Ρωσία ε, έναντι των τρίτων χωρών όπως η Ουκρανία θα πρέπει να εγκριθούν από την Ευρασιατική Ένωση και όχι μόνο από τη Ρωσία πλέον. Σε ποιο βαθμό λοιπόν η Λευκορωσία και το Καζακστάν πρόκειται να ακολουθήσουν την ρωσική γραμμή είναι καθοριστικό. Κάτι άλλο που είναι επίσης καθοριστικό και είναι ιδιαίτερα πολιτικού χαρακτήρα είναι η μη δημοκρατική ε, τάση όλων των μελών της Ευρασιατικής Ένωσης με πολύ χαμηλό επίπεδο κράτους δικαίου. Αυτό αφήνει μεγάλο περιθώριο ελιγμών όταν υπάρχουν συζητήσεις λόγω χάρη μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας. Οι δασμοί για την Ουκρανία θα πρέπει να αυξηθούν ή όχι. Ε, έτσι δεν υπάρχει ευθυγράμμιση μόνο με το τι λέει η Ρωσία, αλλά και με τη Λευκορωσία και, την, ε, και το Καζακστάν που ερμηνεύουν το τι συμβαίνει με την Ανατολική γειτονία. Το τι συμβαίνει τώρα σε επίπεδο του, ε, της, στο επίπεδο της Ρωσίας οι διεθνείς επιστήμονες από την εξή άποψη. Κατά πόσον στην ευρωσιακό χώρο μπορεί να υπάρξει βαθύτερη ένωση εξαρτάται από το κατά πόσον η Ρωσία θα είναι και ένας καλός εταίρος. Το είδαμε και από τον Νοέμβριο ε, με την επίσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και οι Λευκορώσοι και οι Καζάκοι είπαν ότι είμαστε ισότιμοι εταίροι σε αυτήν την ένωση. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ενίσχυση αυτής της ένωσης, η Ρωσία προσπαθεί να έχει μια πολυμερή προσέγγιση, αλλά τα πράγματα αλλάζουν όταν πρόκειται για διεύρυνση της ένωσης αυτής. Ήδη από τον τρόπο με τον οποίο προσεκλήθη να συμμετάσχει στην Ευρασιατική Τελωνική Ένωση Λευκορωσία, το είδαμε αυτό. Αλλά και από την απόφαση του Σεπτεμβρίου την απόφαση της 3ης Σεπτεμβρίου, όπου μονομερός και απροσδόκητα ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Αρμενία θα συμμετάσχει στην ε, ε, Τελωνιακή Ένωση. Ξέρουμε ότι έγινε μία μόνο συνάντηση και υπήρξε ένα συγκεκριμένο είδος επιχειρημάτων. στο ό,τι λοιπόν αφορά την διεύρυνση της Ευρασιατικής Ένωσης, είναι ένα εγχείρημα μόνον της Ρωσίας. Η Λευκορωσία και το Καζακστάν έχουν πει ελάχιστα σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά του προ την Ουκρανία ή την Αρμενία. Εντό λοιπόν του ευρασιατικού καθεστώτο είναι πολύ λιγότερο πολυμερή η Ρωσία από ό,τι ήταν ε, ενεργή εκτό του ευρασιατικου καθεστωτος ειναι πολυ λιγοτερο πολυμερης αυτό. εκτο του πλαισιου αυτο ομως το 2011 ο, κύριος, ο πρόεδρο Πούτιν εξέφρασε την ε, πεποίθηση του ότι μπορεί να εμπιστευτεί τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, τη Λευκορωσία και το Καζακστάν και εφόσον υπάρξει ανάγκη να κλείσουν τα σύνορα με την Ουκρανία λόγου χάρη, ε, η Λευκορωσία και το Καζακστάν θα συμφωνήσουν. Δεν φαντάστηκε λοιπόν, δεν φανταζόταν ότι μπορεί να υπάρξουν αντιρρήσει. Αυτό που λέει και η διαφάνεια ω τελευταίο σημείο είναι ότι η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλά εργαλεία και πολυμερή και διμερή για να επηρεάσει για να επηρεάσει τους ανατολικούς της το τελευταίο από αυτά είναι η συμφωνία CIS του 2011 που επιτρέπει σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε επίθεση προς τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιηθούν ε, δραστικά μέτρα. είναι πολύ ευρία διατύπωση αυτή. Η Ρωσία έχει ήδη πει ότι θα κάνει χρήση της δυνατότητας της συγκεκριμένης. Πολύ σύντομα τώρα, η μόνη χώρα που... Ε, μάλλον οι χώρες που μπορούν ε, να, προσελκύσουν, μπορούν να ε, ε, προσελκύονται προς αυτήν την Ένωση και η μόνη χώρα που προσελκύθηκε ουσιαστικά προς αυτή την Ένωση ήταν η Ουκρανία. Υπήρχαν πολλά οικονομικά ωφέλη και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Εδώ έπρεπε να υπάρξει και μία τεχνική και διοικητική σύγκληση Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά υπήρχε και το πολιτικό επιχείρημα ότι η Ρωσία θα είναι ένας πολύ ισχυρότερο εταίρος έτσι, έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον συμπαρταχθεί λοιπόν κανείς με τη Ρωσία ε, έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έδινε στη χώρα πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Η Ρωσία όμως είναι γνωστή αυτό το είδαμε και από την εκστρατεία στην Ουκρανία, είναι γνωστή για τη χρήση του μπαστούνιου και του καρότου αυτή τη πολιτική, με τα δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία θα έπαιρνε η Ουκρανία τα επόμενα χρόνια. Όμως η Ρωσία δεν προσφέρει μόνο καρότα. Είδαμε και την κίνηση προς, ε, προς το ραβδί που χρησιμοποιεί η Ρωσία στην πολιτική της. Στο πρώτο σημείο το βλέπουμε αυτό και είδαμε και τις εξελίξεις στην Κρυμαία. Αλλά το χαρτοφυλάκιο των μέτρων που μπορεί να επιβάλλει η Ρωσία μπορεί να ενεργοποιηθούν ανά πάσα στιγμή και κατά την άποψή μου θα ενεργοποιηθούν, όπως με οικονομικές κυρώσεις ή με κάποιες ε, μη, μη μέτρα προστασίας, με δασμολογικές ε, αυξήσεις ή με τελωνιακούς ελέγχους ή με αύξηση των δασμών σε επίπεδο αντι-dumping ή με την ενεργειακή διπλωματία της. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό και ε, δυσκολεύει την μετανάστευση των εργαζομένων. Εδώ πρέπει να επικεντρωθούμε και σε αυτό, διότι ότι η πολιτική έναντι μεμονωμένων χωρών μπορεί να μην είναι σημαντική, αλλά όταν συνδυαστούν όλα αυτά τα μέτρα μπορεί να ε, προκαλέσουν ε, σοβαρά προβλήματα στους ανατολικούς εταίρους. Πολύ σύντομα λοιπόν, ε, μικρή παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στη Γεωργία, αυτό που βλέπουμε στη φωτογραφία. Θέλουν να μπορούν να εξάγουν και στην ευρωπαϊκή αγορά οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά όταν μιλάμε για τιμωρία, ξέρουμε ότι έχει γίνει στην Μολδαβία με τα εινοπνευματόδη λόγου χάρη. 28% των εξαγωγών της ε, Μολδαβίας κατευθύνονται στην Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανοίξει την αγορά της με το θέμα των ε, σημάτων και των πόρων. Είναι πολύ ανταγωνιστική αγορά βέβαια της Ευρώπης, αλλά η Μολδαβία θα δυσκολευτεί πολύ να δυσδύσει σε αυτή την αγορά. Ενώ τα γεωργιανά και τα μολδαβιανά κρασιά στην Ρωσία χαίρουν μεγάλη εκτίμηση και είναι και πολύ γνωστά. Ε, Όμω υπάρχει και η τιμή τη ενέργεια στη Μολδαβία. Ε, αυτή η αυξητική τάση συνεχίζεται και υπάρχει ένα τεράστιο ενεργειακό χρέο. Και εκεί η Ρωσία παίζει μεγάλο ρόλο. Είναι περίπου 4 δις ε, ευρώ το χρέος της Μολδαβίας για την ε, χρήση φυσικού αερίου και είναι υπεύθυνη για το αέριο της υπερδνηστερίας, για το οποίο δεν έχει κανέναν έλεγχο, ούτε καμία ε, δυνατότητα επιρροής, αλλά και για την μετανάστευση εργαζομένων. Είναι μεγάλες οι ε, μετακινήσεις εργαζομένων μέχρι και 500.000 ανθρώπους και 8 έως 25% του ΑΕΠ. Οι Μολδαβοί λένε 8%, αυτό λένε οι μολδαβικές πηγές, ενώ οι Ρώσοι λένε ότι το 25% του ΑΕΠ της Μολδαβίας προέρχεται από τη μετανάστευση εργαζομένων. Για τη Γεωργία τώρα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά ενώ είναι γείτον της Ρωσίας άμεσα και έχει κοινά σύνορα, έχει καταφέρει να ε, διαφοροποιήσει τις εμπορικές της ε, συνελλαγές ελπίζει να εξάγει περισσότερο στην ε, Ευρώπη από ότι η Μολδαβία, αλλά με το κρασί τα έχει καταφέρει εδώ και δεκαετίας. έχει καταφέρει να πείσει τους Ρώσους καταναλωτές με γλυκά κρασιά και ιδίως όταν, ε, μπόρεσε, όταν υπήρξε η άρξη του εμπάργου ε, του κρασιού στην Ρωσία. Υπάρχει λοιπόν διαφοροποίηση, αλλά παρόλα αυτά είναι ακόμη ευάλωτη και η γεωργία και η μετανάστευση των εργαζομένων μπορεί να γίνει μια απειλή για τη γεωργία. Αλλά ας δούμε την Ουκρανία τώρα. Η Ουκρανία είναι πλέον ευάλωτη χώρα. Λέγαμε ότι η Μολδαβία είναι η φτωχότερη χώρα, αλλά δεν είναι αυτό το μόνο που μετράει. Πώς μπορεί να τιμωρήσει η Ρωσία την Ουκρανία. Ας δούμε τι γίνεται με τις εισαγωγές των σιδηροδρομικών εξοπλισμών. Ξέρουμε ότι ήδη έχει πάυσει τις ε, ε, παραγγελίες της η Ρωσία και μάλιστα εδώ μιλάμε για το 8% των εξαγωγών της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως προς τα μηχανήματα που εξάγει η Ουκρανία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εργοστάσια αυτά βρίσκονται κυρίως στην νότια και ανατολική Ουκρανία. Γι' αυτό λέει η Ρωσία ότι όταν θα κλείσει τα σύνορά της ε, θα είναι πολύ ε, θα δυσχεράνει αυτό πολύ την Ουκρανική ε, οικονομία αλλά και το, εμπάργο, το εμπορικό εμπάργκο σε συγκεκριμένα προϊόντα όπως η σοκολάτα, τα γαλακτοκομικά ή το χείριο, εδώ αυτό μπορεί να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Και με τους τελωνιακούς ελέγχους, βλέπετε τον εμπορικό πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας του περασμένου Αυγούστου. Δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες από τη Ρωσία για το λόγο για τον οποίο τα ουκρανικά προϊόντα δεν μπορούσαν να διασχίσουν τα σύνορα και να φτάσουν στη Ρωσία. Η Ρωσία απλώς χρησιμοποιούσε του τελωνιακού ελέγχου όπω του επέβαλε η Βρασιατική Επιτροπή. Δεν υπήρχαν λοιπόν πολλά που μπορούσε να κάνει η Ουκρανία από νομοθετική άποψη πέρα από το να προσφύγει στον ε, ΠΟΕ. Όμω δεν ήταν και πολύ σαφή τα αίτια. Το κλείσιμο λοιπόν των συνόρων είναι μια διαρκή απειλή με γενικόλογε και σαφεί δηλώσει βλέπουμε να υπάρχουν δασμοί που αγγίζουν τα επίπεδα του αντι-dumping, κάτι μπορεί να παραβιάζει τι δεσμεύσει ε, ως προς τους κανόνες του ΠΟΕ και εδώ είναι πολύ σημαντικό και το κράτος δικαίου. Θα μπορούσα να δώσω συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία αν σα ενδιαφέρουν. Τώρα, το πλέον σημαντικό ίσως από οικονομικής σκοπιάς, το πλέον οικονομικό στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει την Ουκρανία από την πλευρά της Ρωσίας είναι η τιμή της ενέργειας. Αυτό πλήττει την οικονομία της Ουκρανίας σε όλα τα επίπεδα και ξέρουμε ότι η ενέργεια πρόκειται να αυξηθεί. Αλλά και η μετανάστευση των εργαζομένων, κυρίως από τη Δυτική Ουκρανία, όπου οι πολίτες είναι πιο αποφασισμένοι να ε, υποστούν τη ζημιά ε, οι τελευταίες δύο διαφάνειες τώρα είναι σημαντικό ε, το τι ε, λέει η Ρωσία, τι προάγει στις εκφράσεις της και για βραχυπρόθεσμες ε, τιμωρίες και αντίπεινα και για το πώς η Ρωσία μπορεί να χειριστεί μεμονωμένα τις χώρες με συγκεκριμένους συμμάχους της στο εσωτερικό των χωρών η Ρωσία ε, βασίζει την πολιτική της στο συνδυασμό αρνητικών και θετικών μέτρων, όχι μόνο για να προσελκύσει νέα μέλη όπως η, Αρμανία, η Αρμενία, αλλά και να τιμωρήσει αυτούς που απομακρύνονται από τη Ρωσία. Η Ρωσία λοιπόν μπορεί γιατί έχει πολύ μεγάλο κύρο ε, έναντι των ανατολικών εταίρων, μπορεί να επιβάλλει κυρώσει για την απομάκρυνση κάποιων και γι' αυτό θα αυξήσει και το κόστος και τον κίνδυνο εφόσον κάποιοι έχουν στενότερη σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο μια βραχυπρόθεσμη ε, αντιπαλότητα αλλά πρόκειται για εκδίπλωση μακροπρόθεσμης πολιτικής με την πρόθεση να υπονομευτεί η ευρωπαϊκή επιλογή των ανατολικών εταίρων. Δεν τίθεται λοιπόν πλέον θέμα έλξης και προσέλκυσης, αλλά τιμωρίας και μπλοκαρίσματος. Θα κλείσω εδώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Your conclusion has been a ε, το συμπέρασμά σας αποτέλεσε ένα συμπέρασμα που προκαλεί έκπληξη μεγάλη σε όλους. Να δώσω το λόγο, στο, λόγο στον Dr. Κέσσερ από το ε, Πανεπιστήμιο των Βρυξελών. Έχετε το λόγο και θα ήθελα πάλι να προσπαθήσουμε να περιοριστούμε στα 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι κρίσεις που είδαμε στην Ουκρανία τις τελευταίες 10 ημέρες δεν αποτελούν μια νέα πρόκληση απαραίτητα. Πρόκειται για μια κρίση η οποία συνεχίζεται εδώ και πολλά χρόνια, αλλά και πέρασε σε ένα καινούριο επίπεδο. Έχει κλιμακωθεί σε σημείο που κανείς δεν είχε φανταστεί. Περνάμε από έναν ανταγωνισμό, ο οποίος ήταν ε, ένας ανταγωνισμός οικονομικών μέσων. Η Ρωσία που χρησιμοποιούσε ως απειλή κάποια μέτρα περιοριστικά για το εμπόριο, σε ένα de facto ε, ε, προσάρτηση της Κρυμαίας. Και αυτό συνάδει με την πολιτική της Ρωσίας των τελευταίων ετών, αλλά το περνάει αυτό σε ένα νέο επίπεδο, γιατί η Ουκρανία ήταν πάντα ένα σύνορο το οποίο δεν μπορούσαμε να υπερβούμε και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο ενδεχόμενος κίνδυνος που συνοδεύει αυτή την εξέλιξη και δημιουργείται έτσι ένα καινούριο πλαίσιο για την ανατολική γειτονία. Τώρα η συμφωνία σύνδεσης και η υπογραφή της ενδεχομένως να συνοδευτεί όχι από εμπορικά πλέον αντίπεινα, αλλά από στρατιωτικά αντίπεινα. Αυτό είναι καινούριο πλαίσιο λοιπόν. Και πώς διαμορφώνονται λοιπόν οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Να σας πω δύο ιστορίες. Μία σύντομη ιστορία για τα τρέχοντα γεγονότα και μία πιο μακροπρόθεσμη ιστορία για το πώς έχουν εξελιχθεί οι σχέσεις Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια και φυσικά πολλά θα εξαρτηθούν από τις επόμενες εβδομάδες, από τους επόμενους μήνες κατά πόσο θα διατηρηθεί το status quo, ιδιαίτερα τώρα μετά την διενέργεια του δημοψηφίσματος στην Κρυμαία ή κατά πόσο θα υπάρχει περαιτέρω κλιμάκωση ή ενδεχομένως πιο απίθανο αποκλιμάκωση της κατάστασης. Ξεκινώντας με την ε, βραχυπρόθεσμη ιστορία. Τι συμβαίνει σήμερα στην Κρυμαία. Νομίζω ότι de facto εισβολή, προσάρτηση της Κρυμαίας και η υποστήριξη της Ρωσίας στο δημοψήφισμα καταδεικνύουν ότι η Ρωσία έχει ξεπεράσει ε, ε, μια, ένα όριο και έχει δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο και επίσης παραβιάζει πολλές διεθνείς συμβάσεις του ΟΗΕ, του σχετικού χάρτη, ε, του μνημονίου της Βουδαπέσης, του άρθρου 3 του συντάγματος της Ουκρανίας και είναι ασφαλώς πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το παιχνίδι, η αστάθεια της αλλαγής των συνόρων. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα πηγαίνουν και παραπάνω, είναι και παράνομο υπό την έννοια ότι πρόκειται για ένα δημοψήφισμα το ο οποίο δημιουργεί αστάθεια υπό την απειλή των όπλων ουσιαστικά. Η φαρπαγή ε, και προσάρτηση de facto. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει αποδεκτό στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει περιθώριο αλλαγή συνόρων χωρίς να προκύψει μια μακροπρόθεσμη διαδικασία ε, διαπραγματεύσεων. Επίσης, ε, τίθεται και ένα θέμα των προβλημάτων των μειονοτήτων στην Ευρώπη. Έγινε μια αναφορά στην Ανατολική Ευρώπη για, ως μια περιοχή ε, με πάρα πολύ μεγάλη πολυμορφία και τα προβλήματα λοιπόν των μειονοτήτων στην Ουκρανία δεν μπορούν να επιληθούν γιατί η επίλυση του θα σήμαινε ότι θα δημιουργηθούν νέα προβλήματα για τι μειονότητε. Να σα δώσω λοιπόν και κάποιου καινούριου λόγου για την παρέμβαση τη Ρωσία που δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την ευαισθησία για τι ρωσόφωνε μειονότητε, όπω αναφέρεται στον τύπο. Είναι μια δικαιολογία αυτή για στρατηγικού λόγου, ασφαλώ. Η Ουκρανία είναι εξαιρετική σημασία για τη Ρωσία θεωρείται γεωπολιτικός πως από τη Μόσχα ως μια ενδιάμεση ζώνη και το καθεστώς στο Κίεβο που θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο προσάρτηση στο ΝΑΤΟ είναι κάτι το προσχώρηση στο ΝΑΤΟ είναι κάτι το παράδεκτο και φυσικά τίθεται και το θέμα της Κρυμαίας όλος ιδιαίτερος και του αυξήνου πόντου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς κινητοποιεί τις πολιτικές ταυτότητες η Ρωσία στην Ουκρανία για πολιτικούς σκοπούς, αν και συμβαίνει αυτό και αντίστροφα από την Ουκρανία. Με ένα σπάρο τριγώνια θέλει αυτό να πετύχει η Ρωσία μιλώντας για την προστασία των ρωσόφωνων μειονοτήτων, δημιουργεί έτσι μια στρατηγική δικαιολογία και παράλληλα ε, υψώνει το λάβρο της σημαίας για τους Ρώσους πολίτες. Και στο παρελθόν ήταν μάλλον μικρή κινητοποίηση των ρωσόφωνων μειονοτήτων. Δεν ήταν ότι υπήρχε μεγάλη τέτοια ιδέα προσάρτηση στην μητέρα Ρωσία. Και τώρα η εθνοτική μειονότητα που συνέχεια ακούμε στον τύπο είναι κάτι τώρα σαφές. Η Ουκρανία λοιπόν πρέπει να πούμε ότι χαρακτηρίζεται από πολλές μειονότητες που χρησιμοποιούν πολλές γλώσσες, άρα ακόμα και η ρωσική μειονότητα ως ορισμός, ως έννοια είναι κάτι δύσκολο να το αντιληφθούμε. Η στρατηγική λόγη λοιπόν τώρα για τη Ρωσία. Να σας ε, παρουσιάσω τη δεύτερη, τη μακροπρόθεσμη ιστορία. Και αυτή η ιστορία ουσιαστικά έχει να κάνει με τις στρατηγικές ανησυχίες της Ρωσίας. Βλέπουμε ότι υπήρχαν βαθιά δομικά προβλήματα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας και Ρωσίας και Δύσης γενικότερα επί σειρά ετών. Και νομίζω ότι θα είναι σωστό και απαραίτητο αυτά μακροπρόθεσμα να αντιμετωπιστούν προκειμένου να μην καταλήξουν ε, σε σύγκρουση. Να πω δύο λόγια για τη φύση της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας. Ε, κοιτώντας τις ενέργειες ε, του τελευταίου έτους, η πολιτική αυτή χαρακτηρίζεται από μια πολιτική άσκησης μειών και προ προβολής μιας ε, εικόνας ε, εξουσίας, αλλά ουσιαστικά η εξωτερική πολιτική της Ρωσίας ε, διέπεται από το φόβο της ταπείνωσης, γιατί βλέπουμε ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει μειωθεί, έχει συρρυκνωθεί αυτή η πολιτική εξουσία στο παγκόσμιο προσκήνιο και αυτό συνεργατεύεται και από γεωπολιτικές σχετικές πράξεις. Βρίσκεται λοιπόν αρκετά απομονωμένη η Ρωσία και δεν έχει αναγνωριστεί ως, ε, θεωρεί τουλάχιστον, ως μεγάλος παίκτη στο διεθνές προσκήνιο και στην Ευρώπη. Και αυτό έχει κινητοποιήσει και έχει δώσει τροφή σε ε, την αντίληψη ότι υπάρχει αντιρωσική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι αναπτύσσεται μια λογική γεωπολιτικού ανταγωνισμού Ξεκινάμε με το έτος 1999 στην ε, ε, παρέμβαση στο Κωσυφοπέδιο, το οποίο όλος ε, περιέργως έχει αντιστρέψει τώρα η ρωσική πολιτική και χρησιμοποιείται ως επιχείρημα και με την διεύρυνση του ΝΑΤΟ το ίδιο έτος σύζευξη της πολιτικής ευρωπαϊκής γειτονίας και της πολιτικής της Ρωσίας ήταν απόφαση της Ρωσίας να μην συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Έγιναν λοιπόν κάποιες επιλογές και από τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Το 2004 ενισχύθηκε ο ανταγωνισμός αυτός από την Πορτοκαλή Επανάσταση και από τις υπόλοιπες επαναστάσεις που θεωρήθηκε από τη Μόσχα ότι κινητοποιήθηκε και ε, υποδαβλίστηκε από τη βετική πολιτική και από την χώρια, την ιστορική πολιτική και τελικά κλιμακώθηκε στην πολιτική γειτονίας και στη σχετική ε, υπογραφή συμφωνιών σύνδεσης με τις χώρες της πολιτικής σύνδεσης. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε μια λογική ανταγωνισμού. Υποσυνείδητα ενδεχομένως σε μεγάλο βαθμό και βρεθήκαμε σε μια κατάσταση εναλλακτική ε, μάλλον σε μια λογική πολιτικών που αποκλείουν ε, κάποιες χώρες και αυτό δημιουργεί λοιπόν διχασμό στην Ευρώπη και είναι κακό για τις σχέσεις γειτονίας, γιατί χρειαζόμαστε καλές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύγκρουση λοιπόν έχει περάσει σε ένα νέο επίπεδο, σε ένα στρατιωτικό επίπεδο. Αυτές οι επιλογές έχουν γίνει πιο βαθιές και ανακύπτει λοιπόν το θέμα του ρόλου και της θέσης της ε, Ρωσίας στην Ευρώπη ανακύπτει το θέμα των διαχωριστικών γραμμών στην Ευρώπη. Αυτό βράχει μακροπρόθεσμα μετά την ε, κρίση θα πρέπει να τεθεί επιτάπητο στην περίοδο μετά τον Πούτιν και μακροπρόθεσμα θα πρέπει να σκεφτούμε μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Αυτό θεωρώ ότι απασχολεί πολύ τη Ρωσία για να μην πηγαίνουμε από τη μία σύγκρουση στην άλλη. όταν αναφέρθηκε ότι η Ρωσία ανησυχεί, για παράδειγμα, για την πολιτική γειτονία και ότι θεωρείται αυτό απόπειρα επέκταση τη σφαίρα επιρροή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό πραγματικά αποτελεί ένα αληθινό φόβο και ίσω θα πρέπει να αναφερθούμε και, να αντιμετωπίσουμε και το γεγονό ότι δεν έχουμε ευρωπαϊκέ δομέ για να αντιμετωπίζουμε τέτοια θέματα. Ίσως λείπουν κάποιε τέτοιε υποδομέ που θα μα επέτρεπαν να προλάβουμε την ε, εμφάνιση τέτοιων κρίσεων και εδώ και καιρό ζητώ να ε, συμμετάσχει πιο πολύ η Ρωσία. Ίσως χάσαμε στη δεκαετία του 90 την όλη ορμή, την ορμή να αναπτύξουμε ευρωπαϊκές συνολικές ε, δομές που θα επέτρεπαν τη συμμετοχή της Ρωσίας. Τι σημαίνει αυτό στο παρόν συγκείμενο και εδώ πέρα συνενώνονται αυτές οι δύο ιστορίες. Καταρχάς είναι σαφές νομίζω μετά την Κρυμαία ότι οι κυρώσεις είναι κάτι τον αναπόφευκτο και είναι καλό θεωρώ να εισαχθούν σταδιακά προκειμένου να έχει τα περιθώρια η Ρωσία να κάνει ένα βήμα προς τα πίσω, να επαναχωρήσει σε περίπτωση που το επιθυμεί. Και είναι σημαντικό λοιπόν να μην ε, υποτιμήσουμε την ε, οικονομία της Ρωσίας, η οποία είναι περίπου στο μέγεθος της Ιταλίας. Είναι απομονωμένη. υποστηρίζετε, θέλει την υποστηρίξη των άλλων ε, μέλων της ε, ε, Τελωνιακής Ένωσης και θεωρώ ότι θέματα, ε, τα θέματα ενεργειακής εξάρτησης και αυτά ε, υπερτιμούνται. Κοιτώντα αριθμητικά στοιχεία σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι πιο μικρό από, τον, από τα επίπεδα σε απόλυτες τιμές του 1991. Σήμερα λοιπόν έχει περιοριστεί στο 1 τρίτο περίπου, στο 1 τέταρτο σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο που καταναλώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Ρωσία. Σημαντικό ποσοστό, αλλά πιο χαμηλό από αυτό που πολλές φορές ε, προβάλλεται. Νομίζω ότι οι κυρώσεις αυτές ενδεχομένως θα πρέπει να ε, συνδεθούν και με κάποιες μακροπρόθεσμες ε, υποσχέσεις. Κάνει ένα βήμα πίσω η Ρωσία και σε περίπτωση που υπηρεθεί η κρίση. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Αυτή η μακροπρόθεσμη προοπτική, γιατί η μπορεί να υπάρξει νέα κλιμάκωση. Αν θέλουμε λοιπόν να αποφύγουμε νέες συγκρούσεις στο μέλλον, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Ανατολική Ευρώπη δεν είναι η Ρωσία μόνο. Και αυτό τι σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις ε, Ανησυχίε τη Ρωσία για τι ρωσόφωνε μειονότητες, ενδεχομένω, να πρέπει να συζητήσουμε και θέματα εξωτερική πολιτική τη Ουκρανία σε μετέπειτα στάδιο και να συζητήσουμε και το ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα η Ουκρανία για την Ανατολική Γειτονία συγκεκριμένα. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τη Συμφωνία σύνδεση και το θέμα του ε, ελεύθερου και βαθιού συνεκτικού εμπορίου είναι ένα θέμα που έχει αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την προσχώρηση κάποιων χωρών στην ε, σφαίρα οικονομικής επιρροής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να συμμετάσχει η Ρωσία αν θέλουμε να ε, εξέλθουμε της κρίσεις, και θα πρέπει αυτός ο νέος παράγοντας που είναι ο διχασμός της Ευρώπης σε δύο τμήματα ε, η Ανατολική Γειτονία και η Τελωνιακή Ένωση θα πρέπει να προσεγγίσουν τα δύο αυτά τα στοιχεία το ένα το άλλο για να κινηθούμε προς ένα χώρο ελεύθερου εμπορίου. Κατανοώ ωστόσο ότι αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα καθήκοντα τα οποία ενδεχομένω να φαντάσουν και αδύνατα σε αυτή τη φάση. Αν θέλουμε όμως, επαναλαμβάνω, να αποφύγουμε ένα σενάριο όπου θα κινούμαστε από τη μία κρίση στην άλλη, θα πρέπει να κοιτάξουμε και αυτή τη μακροπρόθεσμη διάσταση. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Βίγκαν τώρα, διευθυντής ε, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Έχετε το λόγο κύριε Βίγκαντ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τους διοργανωτές αυτής της δημόσιας ακρόασης ε, που είναι τόσο επίκαιρη γιατί το θέμα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. Ελπίζω να έχουμε αποκλιμάκωση τις επόμενες μέρες και σίγουρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΔΑ καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για την αποκλιμάκωση αυτή και ελπίζω η Ρωσική Συνομοσπονδία να ανταποκριθεί σε αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα το Συμβούλιο της το μόνιμο Συμβούλιο της ΟΑΣΕ στη Βιέννη θα λάβει πολύ σημαντικές αποφάσεις και δεν αποκλείεται στο άμεσο μέλλον τις επόμενες μέρες ε, να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για την ε, αποστολή αντιπροσωπείας παρακολούθησης στην Ουκρανία που θα είναι ένα πολύ καλό πρώτο σημάδι ε, σε μια διαδικασία αποκλιμάκωσης. Δεν ξέρουμε τι θα πει αύριο ο κύριος Πούτιν στην ειδική του ομιλία προς την Ντούμα για την κατάσταση της Κρυμαίας. Οι εξαγγελίες του θα μπορούσαν να έχουν Πολύ πλούσιο περιεχόμενο. Ελπίζω πάντως ε, να αποφύγει η Ρωσία να προσαρτήσει τμήμα τρίτης ε, χώρας. Γιατί κάτι τέτοιο είναι παράνομο, αθέμητο και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και μάλιστα και της χάρτας των Ηνωμένων για να μιλήσουμε για τις διμερείς συμφωνίες της Ρωσίας ε, με την Ουκρανία. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, έχουμε δυστυχώς ε, κάποιες ε, αρνητικές εξελίξεις. Περάσαμε δηλαδή από διάφορες προφορές οικονομικής ολοκλήρωσης ε, σε ανοιχτή πολιτική αντιπαράθεση με σημαντικές επιπτώσεις και στο θέμα της ασφάλειας. Και για πρώτη φορά, μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, έχουμε πια ανοιχτές προκλήσεις την τελική πράξη του Ελσίνκη. Γιατί εκεί εδώ βλέπουμε πια να αμφισβητείται η αρχή της εδαφικής ακεραιότητας. Και επαφείεται ε, η αλλαγή των συνόρων σε μονομερή απόφαση χωρών μελών. Και αυτό είναι μια νέα κατάσταση που χρήζει πολύ σοβαρής ε, αντιμετώπισης. Ο συνάδελφο Μπάλα από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μιλήσει περισσότερο για το ιστορικό τη κατάσταση και τι συγκεκριμένε οικονομικέ προκλήσει. Αλλά εγώ διαφωνώ με, την, με τον προηγούμενο ισχυρισμό ότι όλα αυτά προκλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφωνώ γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μια μετριοπαθή οικονομική πολιτική προς πολλές τρίτε χώρε και στις χώρες ανατολικής ε, Γειτονία αν και οι συγκεκριμένες συμφωνίες ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξες. Πάντως το λογικό αυτών των συμφωνιών είναι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των μη δασμολογικών φραγμών. Οπότε δεν μειώνονται μόνο οι δασμοί ή καταργούνται οι δασμοί και οι ποσοστώσεις, αλλά ταυτόχρονα εφαρμόζονται οι ίδιοι, οι κανόνες και προδιαγραφές ε, για όλα τα προϊόντα ώστε να κινούνται ελεύθερα από ένα οικονομικό χώρο προς τον άλλο. Ουσιαστικά δηλαδή και de facto εποφελούνται της ε, κατάστασης της μεγάλες παγκόσμιες αγορές. Και κάτι που κάνουμε ε, με άλλες ε, τρίτες χώρες, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε με τις χώρες ανατολικής γειτονίας. Κάτι που είναι απαραίτητο ε, αλλά έχουμε και νέε μορφέ ευρωετική ολοκλήρωση. Και όταν ξεκινήσαμε το 2007 τι διαπραγματεύσει με την Ουκρανία, δεν υπήρχε καμία ένδειξη κάτι τέτοιο. Και το 2003 όταν ξεκίνησε η Ανατολική Πολιτική Γειτονία, ακόμη λιγότερο είχαμε τέτοιε ενδείξει. Όταν ξεκινήσαμε το 2009 την Ανατολική Εταιρική Σχέση, άρχισαν να δημιουργούνται κάποια σημάδια, αλλά ήταν γνω... γνωστή και η φιλοδοξία τη Ουκρανία με διαφορετικές βέβαια πλειοψηφίες και σχετισμούς δυνάμεων στη Ράντα, στην κουρανική Βουλή και μία διάσταση απόψεων και ε, είχαμε ακόμη και έκφραση συμφερόντων από την Ανατολική Ουκρανία και βιομηχάνων από την Ανατολική Ουκρανία που τάσσονταν υπέρ της ε, συμφωνίας με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε για μας από πολιτική άποψη φτάνουμε τώρα στο κύριο πολιτικό θέμα, το σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας των διαφόρων χωρών, όπως εκφράζεται αυτή από δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις και κοινοβούλια. Αυτή λοιπόν, αυτο ο σεβασμός της εθνικής κυριαρχίας ε, θα είναι το... Ο κανόνας ή θα επιστρέψουμε σε παλιά παιχνίδια ε, σφαίρας επιρροής που ήταν ε, χαρακτηριστικά προηγούμενων εποχών, όπως είπε και η Άγγελα Μέρκελ στην ομιλία της περασμένης εβδομάδας στην Bundestag. Είναι σημαντικό θέμα λοιπόν εξωτερικής πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά και πέραν αυτής. Γιατί αν αυτή η προσέγγιση γίνει υπόδειγμα για την διαχείριση εκκρεμών ζητημάτων, τότε αυτό είναι κάτι που όχι μόνο θα επαναληφθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά μπορεί να ε, επαναληφθεί από άλλες χώρες εις βάρος της ε, Ρωσικής Ομοσπονδίας. Από χώρες που έχουν ε, ισχυρό στρατό, για παράδειγμα, στην, σε οποιαδήποτε ζώνη του κόσμου. Γι' αυτό και ήταν στεναρή η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για πρώτη φορά σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων αποφάσισε να εφαρμόσει ε, συγκεκριμένα μέτρα περιοριστικά απέναντι στη Ρωσική Ομοσπονδία. Και έχουμε και νομοθετικά μέτρα και άλλου είδους μέτρα. Ήταν πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το σημάδι που δώσαμε, αυτό το μήνυμα, γιατί ήμασταν ανέκαθεν κατά της έγκρισης και επιβολής κυρώσεων κατά στρατηγικών ε, εταίρων μας, όπως είναι η Ρωσική Ομοσπονδία, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κάτι τέτοιο. Είχαμε και βέβαια την ε, πρόταση για τον κατάλογο Μαγνίτσκι. Βέβαια τώρα έχουμε πολύ πιο σοβαρές προκλήσεις και θα πρέπει και η αντίδρασή μας και η αντιμετώπιση είναι πολύ σοβαρή. Τώρα έχουμε περάσει τη δεύτερη φάση αυτής της αντίδρασης ε, και ελπίζουμε ότι το μήνυμα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων είναι σαφές. Η Ρωσία δεν χρειάζεται μια νέα Κρυμαία. Και αν δεν έχουμε κάποια αποκλιμάτωση, φοβάμαι ότι η αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα περάσουν σε λήψη και νέων μέτρων. Το είπαν και στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου. Και μην ξεχνάμε ότι έπεται νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Παρασκευή και Σάββατο. Η υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ουκρανία και η υπογραφή των πολιτικών διατάξεων κυρίως είναι πολύ χειρό πολιτικό μήνυμα και σε χαλεπούς καιρούς για την Ουκρανία μάλιστα. Η συμφωνία αυτή της τελικής πράξης της Συμφωνίας Σύνδεσης περιλαμβάνει και τη δέσμευση των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων να προχωρήσουν στην ε, υπογραφή του συνόλου της συμφωνίας συμπεριλαμβανομένης και της DCFTA αυτής της σφαιρικής και εις βάθος συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών. Εμεί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν θέλησαμε να δημιουργήσουμε σύστημα σφαιρών επιρροή. Κάτι τέτοιο είναι ξένο προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια τέτοια προσέγγιση. Εμεί πιστεύουμε σε εμπορικά μέτρα και στη δημιουργία νέων επενδυτικών ευκαιριών. Και μάλιστα όταν ο πρόεδρος Γιαννουκόβιτς, ο πρώην πρόεδρο τη Ουκρανίας, μας, έλεγε ότι το 60% της Ουκρανικής βιομηχανίας βρίσκεται σε ρωσικά χέρια, αυτό δεν το, ξε, δεν γνωρίζαμε, δηλαδή ότι η ιδιοκτησία, το 60% της Ουκρανικής βιομηχανίας είναι ρωσική, ε, και αυτές οι επιχειρήσεις θα επωφελούνταν από τη Συμφωνία Σύνδεσης και τη συμφωνία, την Σφαιρική και Βάθος Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Βέβαια τα διοικητικά θέματα ε, θα μας τα εξηγήσει ο συνάδελφος. Θα ήθελα να επισημάνω εδώ ότι η πολιτική μας απέναντι στη Ρωσία την τελευταία δύσκολη αυτή χρονιά χαρακτηρίστηκε αφενός από τον εκφοβισμό των ε, εταίρων μας της ε, Ανατολική εταιρική σχέση εκ μέρους της Ρωσίας. Ε, μας ανέλησε τι διάφορε μορφέ αυτού του εκφοβισμού η Δ. Βόλτσουκ. Εμείς ε, θέλουμε να στηρίξουμε τους εταίρους μας, αλλά εδώ δεν βρισκόμαστε σε διαδικασία σταδιακής ε, αύξηση των εντάσεων με τη Ρωσία. Εμείς θέλουμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις ανατολικής εταιρικής σχέσης, υπογράφοντας συμφωνίες σύνδεση με τις χώρες αυτές, αλλά κάναμε και τεράστιες προσπάθειες οργανωτικές για να καταλήξουμε σε εναρμόνιση κανόνων και προδιαγραφών σε πολλούς τομείς που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ε, επιτυχή ανάπτυξη και νέων βιομηχανικών κλάδων ε, στη Ρωσία και την πρόσβασή τους στις δικές μας αγορές και μάλιστα είχαμε και δάνειο ενός δισεκατομμυρίου ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πέρυσι για προώθηση και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Φέτος έχουμε τη χρονιά της επιστήμης με τη Ρωσία και ε, στηρίξαμε την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ το 2012 και στον ΩΣΑ. Βέβαια, η κατάσταση έχει παγώσει από πολλές απόψεις και τον Ιανουάριο είχαμε σημαντική σύνοδο κορυφής που δεν ήταν μια συνηθισμένη σύνοδος κορυφής εξαιτία των διαφορών που έχουμε ε, και τις, στάσεις, τις διαφορετικές που θέτουμε απέναντι στους γείτονές μας που είναι κοινοί. Και Υπάρχει παράταση για συμφωνία στρατηγική εταιρική σχέση με τη Ρωσία, γιατί έχουμε αλληλεξάρτηση. Και μάλιστα ε, είναι περίεργο που η Ρωσία δίνει περισσότερη έμφαση στις εμπορικές σχέσεις με την Ουκρανία που έχει το 5% των εμπορικών συναλλαγών και όχι με την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει το 50% το εμπορίο και το 80% των αλλαδοπών επενδύσεων. Πάντως πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ευαθύνουμε αυτή τη στρατηγική σχέση με τη Ρωσία και να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία πλαίσιο, ταυτόχρονα αναλύοντα τον αντίκτυπο, τον οικονομικό αντίκτυπο σε πιο επίσημε διαπραγματεύσεις, γιατί είχαμε και άτυπε διαπραγματεύσει με την Ουκρανία για την ρωσική βιομηχανία. Ο συνάδελφος θα το αναφέρει αυτό πιο διεξοδικά, αλλά θα ήθελα να πω ότι η κοινή προοπτική μας είναι να δημιουργήσουμε μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, Τελωνιακής Ένωσης της Ευρασίας. Να δημιουργήσουμε κάτι δηλαδή που ε, δεν περιορίζεται ε, όπως συνήθως στη σχέση με τη Ρωσία, αλλά να δημιουργήσουμε ένα, ένα κοινό οικονομικό χώρο. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει το σεβασμό της Εθνική κυριαρχία των χωρών και τη ελεύθερη επιλογή του για το τι σχέση θα δημιουργήσουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι σχέση θα δημιουργήσουν με τη Ρωσία. Θα θέλουν πιο ε, με μία ζώνη από ό,τι με άλλη, είναι δική του ελεύθερη επιλογή. Δεν θα γίνουν επιβολές όπως συνέβη με την απόπειρα της Ρωσίας να επιβάλλει τις επιλογές στην αρμενική κυβέρνηση, στην Ουκρανική. Ευχαριστώ κύριος Μπάλας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Υπόθηκαν πολλά για τις οικονομικές επιπτώσεις και ποινές που μπορεί να επιβάλλει η Ρωσία στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σας πω κάποιες λεπτομέρειες για τη φύση των σχέσεων αυτών και ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των μεν και των δε. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, χώρες δηλαδή, που ήταν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης είχαν ήδη πολύ στενές οικονομικές σχέσεις. Μετά την ε, κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης διατήρησαν αυτές τις σχέσεις και παρέμειναν στο πλαίσιο της Ομοσπονδίας Ανεξαρτήτων Κρατών με στενές με την κοινοπολιτεία ανεξαρτητών κρατών, με στενές σχέσεις μεταξύ των πρώην Σοβιετικών κρατών. Κάτι κατανοητό και από την σκοπιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο το δεχόμαστε και το στηρίζουμε. Η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Ελεύθερων Συναλλαγών της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών με πολυμερή προσέγγιση ισχύει εδώ και 20 χρόνια πλέον. Όμως πρόκειται για μια σχέση που βρίσκεται σε τέλμα. Διότι επί μια εικοσαετία αφορούσε κυρίως τις ε, συναλλαγές και τις, ε, την, το εμπόριο προϊόντων. Άλλοι τομείς δυναμικής οικονομικής συνεργασίας, υπηρεσίες, επενδύσεις δεν καλύπτονται και ελάχιστα τα μη δεσμολογικά μέτρα, που είναι η ε, κύριοι φραγμή αυτή τη στιγμή ε, κατά του εμπορίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιθέτω, εμεί έχουμε αναπτύξει την πολιτική ανατολική γειτονία, αντιδρώντα και αποκρινόμενοι στι ανάγκε των ε, εταίρων μα. Πρώτη πιο μεγάλη χώρα με την οποία αρχίσαμε τις διαπραγματεύσεις και με την οποία είχαμε μια σφαιρική ε, Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου το 2007 ήταν η Ουκρανία. Οι διαπραγματεύσεις αυτές προχώρησαν γρήγορα γιατί από την αρχή ήταν σαφές ότι θα πρόκειται για μια σχέση που θα ξεπερνούσε το ελεύθερο εμπόριο και θα κάλυπτε όλους τους τομείς που προανέφερα προσφέροντας σοβαρές βελτιώσεις στις ε, σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας, στο ευρύτερο πλαίσιό τους. Η ανατολική ε, συνεργασία άρχισε να περιλαμβάνει και άλλες χώρες πέραν της Ουκρανίας με, παρόμοιους, με παρόμοιες αρχές και στόχους όπως αυτοί που τέθηκαν το 2007. Είδαμε άλλους πέντε πιθανούς ανατολικούς εταίρους πέραν της Ουκρανίας και ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις με τρεις από αυτές, Μολδαβία, Γεωργία και Αρμενία. Δύο μήνες μετά την απόφαση του 2009 της άνοιξης του 2009 για την δημιουργία της, των πολιτικών αλατολικής γειτονίας ε, υπήρξε μια ξαφνική αλλαγή. Τον Ιούνιο του 2009 η Ρωσία και άλλες δύο χώρες, η Λευκορωσία και το Καζακστάν, αποφάσισαν να ξεκινήσουν τη δική τους τελωνιακή ένωση ε, μεταξύ των τριών, μία στενότερη δηλαδή και βαθύτερη οικονομική σχέση μεταξύ των τριών αυτών χωρών. Περισσότερο από ό,τι στο πλαίσιο τη κοινοπολιτεία ανεξαρτητών κρατών. Όμω υπάρχει μια καθοριστική διαφορά μεταξύ τη προσέγγιση τη προσέγγισης τη Ένωση και τη προσέγγισης που επέλεξε η Ρωσία και που ακολούθησαν οι εταίροι της. η πρόταση για συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και για ελεύθερες εμπορικές σχέσεις επιτρέπει την συμμετοχή πολλών εταίρων. Πολλές εμπορικές συμφωνίες μπορεί να συνεπάρχουν παράλληλα και μία χώρα που συνάπτει μια τέτοια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου έχει το δικαίωμα και την ελευθερία να συνάψει και άλλες ε, σχέσεις με άλλους εταίρους, άλλες συμφωνίες με άλλους εταίρους, με διαφορετικές αλλά συμβατές συνθήκες. Συνολικά λοιπόν η εμπορική κυριαρχία, η εμπορική εθνική κυριαρχία των εμπορικών εταίρων δεν αμφισβητείται. Ενώ η τελογική ένωση είναι κάτι διαφορετικό, είναι μια μονομερής σχέση και τα μέλη μιας τελωνιακής ένωσης από τεχνικής και νομοθετικής πλευράς δεν μπορούν να περάσουν σε ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές με οποιονδήποτε άλλον. Από αυτήν λοιπόν τη σκοπιά συγκυρία της επιλογής να ξεκινήσει αυτή η Τελωνική Ένωση ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα, διότι δύο χρόνια μετά την αρχή των διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ελεύθερο εμπόριο με την Ουκρανία, η Ρωσία αποφασίζει να δημιουργήσει τη δική της Τελωνική Ένωση. Κάτι που εξορισμού σημαίνει ότι η Ουκρανία δεν θα ήταν σε θέση να συμμετάσχει στην Τελωνιακή Ένωση από τη μια, λόγω της φύση ακριβώς της Τελωνιακής Ένωσης που περίγραψα και λόγω των εμπορικών της διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την ευρωπαϊκή τουλάχιστον οπτική γωνία αυτό ήταν ε, μάλλον ένα θλιβερό γεγονός αλλά ε, ενθαρρύνθηκαν ε, οι εταίροι μας της Ανατολικής Γειτονίας να προχωρήσουν στις σχέσεις τους με την Ρωσία και στο πλαίσιο της κοινοπολιτείας ανεξαρτητών κρατών και των σχετικών συμφωνιών αυτό ήταν απόλυτα εφικτό για τις εμπορικές σχέσεις ε, για την ανταλλαγή προϊόντων αλλά και τις υπηρεσίες, τις ε, επενδύσεις και τις δημόσιες προμήθειες δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο. Οι επιλογές αυτές δείχνουν ότι δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά η Ρωσία που άρχισε να βλέπει την οικονομική συνεργασία ως ένα μέσο ανταγωνισμού σε γεωπολιτικό επίπεδο για να κυριαρχήσει ε, στην περιοχή στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας τώρα, πέραν από το γεγονός αυτό και παρά το γεγονός αυτό, η Ρωσία ως πέρσι δεν είχε γύρει σοβαρές αμφιβολίες για τις ε, σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και άλλους εταίρους. Έχουμε στενότατες σχέσεις με τη Ρωσία, ετησίως έχουμε δύο συνόδους κορυφής, κάτι που είναι ε, κάτι καθιερωμένο μεταξύ εμπορικών εταίρων, ε, συστηματικές εμπορικές συνομιλίες, την δεδηλωμένη αντίθεση της Ρωσίας με εμπορικές, για τις εμπορικές συμφωνίες με, τους Ανατολικ, με, την, με τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας, που τώρα όμως ανακαλύπτουμε, γιατί σήμερα δεν είχαμε κανένα τέτοιο δείγμα. Οι διαπραγματεύσεις προχωρούσαν χωρίς σοβαρά προβλήματα. Και με την Ουκρανία ολοκληρώθηκαν στο τέλος του 2011. Τότε ο πρόεδρος Γιαννουκόβιτς εξασκούσε τα καθήκοντά του και σε εκείνη τη χρονική περίοδο δεν υπήρχαν μείζωνα προβλήματα, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζαμε. Τα προβλήματα αυτά ξεκίνησαν μόλις πέρυσι το καλοκαίρι. Ξαφνικά ακούσαμε ότι η Ρωσία αρχίζει να λαμβάνει μέτρα ε, κατά της Ουκρανίας, όχι τόσο πολύ δασμολογικά, διότι η Ρωσία έγινε μέλος του ΠΟΕ, οπότε δεν μπορούσε να υπάρξει πρόβλημα με μη δεσμολογικά μέτρα, αλλά με τεχνικούς φραγμούς, με ε, εντατικούς τελωνιακούς ελέγχους και κάποια άλλα μέτρα, που κατά την άποψή μας ήταν παράνομα από τη σκοπιά του ΠΟΕ, από ένα μέλος του ΠΟΕ, ε, την Ρωσία, προς ένα άλλο επίσης μέλος του ΠΟΕ, την Ουκρανία. Μέτρα παρόμοια με αυτά που ελήφθησαν κατά της ε, Μολδαβίας και της Γεωργίας. Ακούμε διαρκώς ότι τα μέτρα αυτά είναι και δικαιολογημένα και σωστά τεκμηριωμένα. Κατά την άποψή μας όμως ε, υπήρχαν σοβαρές αμφιβολίες και ενδιασμοί για την αιτιολόγηση των μέτρων αυτών τι είδαμε να συμβαίνει στην πράξη. Η ε, ένταση τη ε, εφαρμογή των μέτρων αυτών δυσκόλεψαν, δυσχέραναν πολύ τι οικονομικέ μα σχέσει. Το περασμένο λοιπόν καλοκαίρι, μια σειρά από μέτρα ελήφθησαν κατά τη Ουκρανία και ξέφνη η ουκρανική σοκολάτα βρέθηκε να περιλαμβάνει βλαβερές ουσίες. Οι εισαγωγές της έπρεπε να, να, Το ίδιο και με κάποια τρόφιμα που μέχρι τώρα τότε πολλούνταν στην ρωσική αγορά αποτελούσαν κίνδυνο για την υγεία των Ρώσων καταναλωτών. Τα ουκρανικά προϊόντα ξαφνικά δεν έφταναν στο ύψος των ρωσικών τεχνικών προτύπων. Αυτά ως τον Νοέμβριο, όπου η Ουκρανία αποφάσισε επί Προέδρου Γιαννουκόβιτς να μην υπογράψει την ε, συμφωνία ε, ελεύθερου εμπορίου. Ξαφνικά τα προβλήματα αυτά εξαλείφθησαν. Οι ουκρανικές εξαγωγές αμέσως έγιναν καλής ποιότητας, υγιεινές, τα μέτρα των συνοριακών ελέγχων έπαυσαν και η Ουκρανία ξανάρχισε να εξάγει στη Ρωσία μέχρι το Φεβρουάριο φέτος, όπου τα προβλήματα επανεμφανίστηκαν πήγαμε πάλι πίσω στην κατάσταση του Αυγούστου. Ε, τα ουκρανικά προϊόντα έγιναν και πάλι βλαβερά για τους Ρώσους καταναλωτές. Δεν φαντάζομαι να χρειάζεται να σχολιάσω περαιτέρω για τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία χρησιμοποιεί αυτά τα οικονομικά μέτρα κατά των εταίρων της. Ε, επιτρέψτε μου εντάχει να εξηγήσω τι σημαίνουν όλα αυτά για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Όπως αναφέρθηκε η Ρωσία από τον Αύγουστο του 2012 είναι ε, μέλο του του οργανισμού ε, που ε, την έφερε στα, στην, ε, συμμετοχή τη στον ΠΟΕ. Υπήρξαν πολλά μέτρα απελευθέρωσης, χρησιμοποιήθηκαν πάλι κάποιοι δασμοί αλλά σε έναν περιορισμένο βαθμό, προβλέψαν νέοι κανόνες, αλλά ήταν σαφές από την αρχή ότι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει μέτρα προστατευτικά προστατευτισμού για ευαίσθητους κλάδους όπως η γεωργία, η, τα οχήματα και άλλους κλάδους χρησιμοποιώντας μέτρα και μεθόδους που έχω ήδη αναφέρει στην περίπτωση της Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν εξαναγκάστηκε να κάνει κάτι το ε, άνευ προηγουμένου με την ε, ενεργοποίηση της διαδικασίας επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ. η χρονιά του μέλητος, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, τελικά δεν πήγε καλά, ακριβώς λόγω αυτών των τριγμών. Ε, ο συνάδελφος ανέφερε τη νέα συμφωνία ε, για την εταιρική σχέση και τη συνεργασία που τελικά δεν προχώρησε επί έξι χρόνια αφού ξεκίνησαν οι συνομιλίες, η Ρωσία δεν ήθελε να λάβει καμία επιπλέον δέσμευση στον εμπορικό και οικονομικό χώρο που ουσιαστικά ε, καθορίζει τις σχέσεις μας και για, την... για τους περιβόητους στόχους Λισαβόνα 2 Βλαδιβοστόκ. Θα μας άρεσε πολύ οι προϋποθέσεις αυτές να ισχύσουν, αλλά το πρόβλημα είναι ότι πέραν της πολιτικής διάστασης που έχει προκύψει και προσφάτως, αλλά και από τις οικονομικές, τίποτα δεν έχει προχωρήσει από την πληρωσική πλευρά για να προχωρήσουμε με αυτό το εγχείρημα. Η Ρωσία ε, δυσκολεύει την προσχώρηση ενός άλλου μέλους της Τελωνιακής Ένωσης, του Καζακστάν, με καμία απολύτως μείωση στις δασμολογικές προϋποθέσεις που θα πετούνταν βάσει των κανόνων του ΠΟΕ ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει το Καζακστάν. Η Λευκορωσία απέχει πόρο από την εκπλήρωση των όρων του ΠΟΕ οπότε η Τελωνιακή Ένωση αυτή καθεαυτή δεν συνάδει με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον ΠΟΕ το ελεύθερο εμπόριο ε, Λισαβόνας Βλαδιβοστόκ θα σήμαινε και άνοιγμα της αγοράς. Αυτή τη στιγμή έχουμε σοβαρότητες αμφιβολίες για το κατά πόσον αυτό είναι μια πιθανότητα που μπορεί κάποτε να υλοποιηθεί στη Ρωσία με τις σημερινές συνθήκες. Όμως αν η κατάσταση αλλάξει κυρίως στην πολιτική αρένα και στην οικονομική σφαίρα η ευρωπαϊκή πλευρά θα ήταν ε, ιδιαίτερα ικανοποιημένη να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι Εν ώψη και των όσων μόλις μας αναφέρατε, τονίζεται η ανάγκη να γίνει μια επισταμένη συζήτηση και εντελεχή συζήτηση σε ό,τι αφορά τα μέσα που έχουμε, τα εργαλεία που έχουμε και την αποτελεσματικότητά του σε ό,τι αφορά την ανατολική γειτονία. Η Κρυμαία θεωρώ ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ε, η αραβική άνοιξη για αυτά τα μέσα τη πολιτική γειτονία. και θα πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε το θέμα αυτό όχι μόνο γραφειοκρατικά αλλά και στρατηγικά και πολιτικά πέρα από την αξιολόγηση της σχέσης μας με τη Ρωσία γενικά. Νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο το πρόβλημα είναι ότι η Ρωσία ποτέ δεν έχει πάρει στα σοβαρά την ανεξαρτησία των πρώην σοβιτικών δημοκρατιών. Και κατά κάποιο τρόπο, έστω και ενδόμηχα, έχουμε επιτρέψει στη Ρωσία να έχει αυτό το αίσθημα υπερτερήσε ότι αφορά τις χώρες αυτές. Ε πέρα από τις βαλτικές χώρες. Όλα αυτά λοιπόν που ε, βλέπουμε πέρα από την Κρυμαία και ούτω καθεξής ε, καταδεικνύουν την ανάγκη να γίνει μια τέτοια αλλαγή νοτροπίας. Έχουμε λοιπόν κάποιους συναδέλφους. Η κυρία Ρέτσοβα δεν το λόγο. Έτσι μου λέει η γραμματεία. Αν δεν θέλετε να πάρετε το λόγο, κανένα πρόβλημα. Όχι, έχω κάποιες ερωτήσεις να κάνω. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω βουλγάρικα. Σας παρακαλώ λοιπόν βάλτε τα ακουστικά σας. Э, э, э, μιλήσω για τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών αυτών. Ρωτώ, κατά πόσον οι εμπειρογνώμονές μας, τους οποίους παρεμπιπτόντως ευχαριστώ για την παρουσίαση και τα σχόλια που κάναν, πολύ αξιόλογα. Ρωτώ όμως το εξής, οι σχέσεις ε, με την Ρωσία έχουν διαμορφωθεί σε σωστή βάση από την αρχή της ανατολικής ε, γειτονίας. Ποια είναι η άποψη των εμπειρογνωμών για το εξή. Η αντίδραση της Ρωσίας πώς μπορεί να ερμηνευθεί. Μιλάμε για τις προσδοκίες της Ρωσίας σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αυτή. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι προσδοκίες της Ρωσίας. Μήπως κάτι κάναμε λάθος σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με τη Ρωσία, σε ό,τι αφορά την διάθρωση της Ανατολικής Γειτονίας, μήπως κάτι αμελήσαμε, μήπως κάτι χάσαμε. Αυτό δεν το άκουσα στις ε, ομιλίες, στις παρουσιάσεις. Και ποια είναι η άποψή σας για τα ακραία κόμματα τα οποία δραστηριοποιούνται στην Ικρανία. Κάποια εξ αυτών συμμετέχουν και στην κυβέρνηση και αυτές οι ενέργειες, αυτές οι δράσεις των κομμάτων αυτών καθορίζουν και την οικονομική και τη στρατηγική πολιτική της χώρας. Να μην τις αφήσουμε λοιπόν κατά μέρο αυτές τις διαδικασίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Στάνο, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ομάδα μου πιστεύει ότι οι κυρώσει οι οποίοι ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα σταματήσουν μόνο κάποιους Ρώσους και Ουκρανούς πλούσιους να κάνουν τα ψώνια τους στο Μιλάνο, εκτός μικροφόνο. Ναι, με ακούσατε. Και φυσικά οι μεγάλοι επιχειρηματίες έχουν ήδη μετακινήσει του, τα χρήματά τους. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτό θα είναι η αρχή μόνο μετά από το δημοψήφισμα υπό την απειλή του όπλου ουσιαστικά στην Κρυμία 41% των ε, κατοίκων της Κρυμαίας θέλουν να προσχωρήσουν στη Ρωσία. Αυτό ήταν τα ποσοστά πριν από κάποιο καιρό και τώρα αυτό το ποσοστό πολύ ενδιαφέρον. Έχει φτάσει 97%, 133%, 123% των ε, πολιτών στη Σεβαστούπολη έχουν καταχωρηθεί για να ψηφίσουν. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει επανέλθει ε, μια νοοτροπία επιχειρηματική της δεκαετίας του 1930 και όχι μια ε, νοοτροπία όπως αυτή μετά το ψυχρό πόλεμο. Μία ερώτηση προς το πάνω ωστόσο, κάτι διαφορετικό. Αν υποθέσουμε ότι μπορεί να μπορούμε να σταματήσουμε τη Ρωσία από το να προσαρτήσει και άλλα τμήματα της Ουκρανίας Θεωρώ ότι αυτή η κίνηση θα ενώσει την Ουκρανία με έναν τρόπο ανεπανάληπτο προς μια ευρωατλαντική προσέγγιση, προς μια ευρωατλαντική ε, κατεύθυνση. Άρα ενδεχομένως ε, ο Πούτιν να ενώσει τους Ουκρανούς ότι, και να αποφασίσουν πολλοί Ουκρανοί ότι προτιμούν να ζουν σε μια δημοκρατία παρά σε μια κλεπτοκρατία την οποία υποστηρίζουν ο Γιαννουκόβιτς και ο Πούτιν. Και φοβάμαι το τι θα επακολουθήσει. Ερωτώ λοιπόν το πάνελ πού θα προσπαθήσει να εξωθήσει καταστάσεις με στρατιωτικά μέτρα. Θεωρώ ότι η Μολδαβία και η σχετική οι Κακαβούζοι είχαν σχετικό δημοψήφισμα πριν από κάποιες εβδομάδες. Πρόκειται να το συνεχίσει αυτό το θέμα στην Μολδαβία. Τι γίνεται με την υπερνηστερία, με τη Γεωργία. Θα είναι η Γεωργία μήπως ο επόμενος στόχος, ε, η Αρμενία. όπου έγινε εκφοβισμός για να μην υπογραφεί η Συμφωνία Ελευθερίου Εμπορίου. Πού θα είναι λοιπόν επόμενος, ποιος θα είναι επόμενος στόχος του. Είναι αδύναμη η αντίδραση των της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είναι πιο δυναμική η αντίδραση των ΗΠΑ, μιας και εξαρτώνται λιγότερο από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και τι γίνεται και με το Ιράν. Σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, για παράδειγμα, που πλευράς της ΗΠΑ. Μήπως αυτός είναι ο τρόπος που θα πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Να υπολογίσουμε την σκληρή στάση των Αμερικανών. Και τελευταίο σχόλιο. Θα πρέπει να απλώσουμε το χέρι προς τους άλλους Ρώσους, τους 50.000 Ρώσους που βγήκαν και διαδήλωσαν κατά των επιθέσεων ε, του Πούτιν κατά της Κρυμαίας και της ε, Ουκρανίας. Να θυμόμαστε ότι υπάρχει και μια διαφορετική Ρωσία πέρα από αυτή του Πούτιν. Ευχαριστώ κυρία Κρόμπεργκ. Αν θα θέλατε να τηρήσετε το χρονικό όριο των τριών λεπτών. Yes. Μάλιστα. Δύο παρατηρήσεις έχω και μια συναφή Αναφέρθηκε ότι η εξωτερική πολιτική της Ρωσίας δεν είναι να δείχνει τους μύστης, αλλά περισσότερο να ταπεινώ, ε, ταπεινώνει και να εκμεταλλεύεται δυναμίες. Χωρίς ε, στρατιωτική επέμβαση η Ρωσία θα ταπεινωθεί, γιατί ε, δεν θα ε, συμμετέχει στη G8, ακυρώνεται η, διάσκε... η σύνοδος κορυφής, οπότε πώς θα αποφύγει αυτή την ταπείνωση ε, και πόσο είναι συναφής η εξωτερική της πολιτική και δεν φοβάται την ταπείνωση. Σε ό,τι αφορά τώρα τη θέση της Ρωσίας στην Ευρώπη. Ερωτώ, πώς αντιλαμβάνεται τη θέση της στην Ευρώπη η Ρωσία υπάρχουν κάποιες οροθετικές γραμμές, γιατί μιλήσαμε για οροθετικές γραμμές και πού βάζει η Ρωσία τις οροθετικές γραμμές στο μέλλον, τις διαχωριστικές γραμμές ή που ελπίζει ότι θα δημιουργηθούν αυτές οι διαχωριστικές γραμμές στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Βούλιανιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μερικές ερωτήσεις που φαίνονται περισσότερο ρητορικέ ερωτήσεις, αλλά με απασχολούν εδώ και αρκετό καιρό και παρόλο που είναι ρητορικέ αυτέ οι ερωτήσει, στην ουσία καλό θα ήταν να συζητηθούν και ενδεχομένω και να απαντηθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αναγνωρίσει το παράνομο ε, δημοψήφισμα που μοιάζει με δημοψήφισμα κορέα. Ωραία. Τι σημαίνει όμω αυτό στην πράξη σε σχέση με την κυριαρχία της Ουκρανίας, το σύνολο της ε, επικράτειάς της. Δηλαδή οι πολίτες της Κρυμαίας θα περιληφθούν στην άρση των, περι, των περιορισμών στις θεωρήσεις κτλ. κτλ. Από την άλλη πλευρά, οι ρωσικές βάσεις ε, δεν θα εγκαταλείψουν ουδέποτε την Κρυμαία. Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος που έχει στα σφρένα ε, γνωρίζει ότι είναι κάτι όχι καινούριο, όχι χθεσινό, αλλά κάτι που δημιουργήθηκε πριν από 50 χρόνια. Η βάση, δηλαδή οι ρωσικές βάσεις στην Κρυμαία. Επίσης, ε, πώς θα προχωρήσει η ενταξιακή προοπτική της ε, Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συνθήκες εδαφικής κυριαρχίας που επιτρέπουν παρουσία ρωσικών βάσεων στην επικράτειά της. Τώρα, πέραν των περιορισμών, είπαμε, μιλήσαμε για περιορισμού στι θεωρήσει, τα ταξίδια ή δέσμευση περιακών στοιχείων. Για ποιου όμω θα ισχύσουν όλα αυτά, για όλους όσους ε, ψήφισαν υπέρ μιας ε, Κρυμαίας που θα προσαρτηθεί στη Ρωσία, που θα ενωθεί με τη Ρωσία. Μήπως μια τέτοια πρόταση έρχεται σε αντίφαση με την ιδέα της ε, κυριαρχίας της, της Ουκρανίας ή της Κρυμαίας. Τώρα, τι γίνεται, τι θα γίνει αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κλείσει κανένας τους αγωγούς φυσικού αερίου θα κλείσει κανένα στις τρόφιγγες. Ευχαριστώ κύριο Σεβερίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τους καλεσμένους μας εμπειρογνώμονες. Αν δεν φοβούνται ότι τώρα... Μήπως τώρα διατρέχουμε τον κίνδυνο να γίνουμε εχμάλωτοι της ε, ίδιας της πολιτικής μας, της ρητορικής μας του πολιτικού μας λόγου, γιατί αυτή την αίσθηση έχω ακούγοντας όλες τις συζητήσεις. Φαίνεται να παρακολουθούμε μια διάλεξη ε, ιδεολογικής διαπαιδαγώγησης. Ε, θυμάμαι τα νανικά μου χρόνια στην κομμουνιστική Ρουμανία, όπου όλα που, όσα έλεγε η Σοβιετική Ένωση, όλα όσα ίσχυαν στο Σοβιετικό μπλοκ ήταν ε, α, α, αλήθεια και όλα όσα έλεγε τότε αντίθετο blog ήταν ε, λαθασμένα. Έχουμε, είχαμε μπερδευτεί με το ποιο έχει δίκιο και ποιο άδικο, γιατί εμεί ε, τα μέλη του Σοβιετικού μπλοκ είχαμε πάντα δίκιο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να εμπλακούμε σε αυτή την ε, λογική, αλλά θα πρέπει να κινητοποιήσουμε μέσα και μηχανισμού και πόρου για να ελοπίσουμε του στόχου μα. Και έχω μια ερώτηση προ του εμπειρογνώμονε. Θεωρείτε ότι στον 21ο αιώνα η πολιτική δεν αφορά πια συμφέροντα, και δεν αφορά μόνο την ε, εξουσία ή το συσχετισμό δυνάμεων ή την ισορροπία δυνάμεων. Γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο, όταν ένας παίκτη όπως η το συσχετισμο δυναμεων η την ισορροπια δυναμεων γιατι αν ισχυει κατι τετοιο οταν ενα παικτη οπως η ρωσια δεν ε, θέλει να παίξει με τους κανόνες του παιχνιδιού που κερδισμένοι, μήπως θα μπορούσαμε να αποφύγουμε να παίζουμε το παιχνίδι του μηδενικού αθρίσματος τουλάχιστον. Και με αυτό το υπόβαθρο και αυτή την άποψη Μήπως θα πρέπει εμείς να υπολογίσουμε τα μέσα μας ε, και τη δυνατότητά μας ε, να φέρουμε τη Ρωσία να δεχτεί τις απαιτήσεις μας. Και υπό αυτό το πρίσμα θεωρείται ότι οι κυρώσεις που εξετάζουμε και που εγκρίναμε είναι αρκετά ε, ισχυρές ώστε να αντισταθμίσουν τις, ε, τα ωφέλη ε, που θα αποκομίσει ο Πούτιν από την πολιτική του. Δηλαδή με τις κυρώσεις θα αναρωτηθεί ο Πούτιν, ο Πούτιν μου τι έκανα, πρέπει να υπαναχωρήσω. Ή μήπως πιστεύετε θα πρέπει να αρχίσουμε τη διαπραγμάτευση μιας ουσιαστικής στρατηγικής συμφωνίας που θα μας επιτρέψει να συνεπάρχουμε όλοι κοινά επιδιώκοντας ο καθένας τα συμφέροντά του. η Ρωσία προσπάθησε να, να διαφυλάξει ε, το, τη θέση της ως παγκόσμιας δύναμης σε μία, ε, σε μία τάξη μετά το ψυχρού πολέμου. Αυτό επιδίωξε η Ρωσία, αλλά δεν κατάφερε. Δεν ε, διαφύλαξε αυτό το, αυτή τη θέση. Και αυτό προσπαθεί να κάνει, να ανακτήσει αυτή τη θέση της υπερδύναμης. Αυτό όμω μπορεί να επηρεάσει τα δικά μα συμφέροντα. Οπότε τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κάνουμε. Παρακαλώ. Τρία λεπτά δείχνει ο μιλητή. Ο κ. Μπουτικόφερ, τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κάνουμε για να διαπραγματευτούμε αυτή τη θέση που διεκδικεί η Ρωσία στην σημερινή παγκόσμια τάξη. Ευχαριστώ Ξέρετε ότι ένας καθηγητής διεθνούς δικαίου λέει ότι η μόνη έγκυρη σχολή σκέψης είναι ο πολιτικός ρεαλισμός. Όλοι οι υπόλοιποι παίζουν ουσιαστικά με τις έννοιες. Μόνο ο ρεαλισμός έχει εφαρμογή. Τώρα θα καλέσω τους προσκεκλημένους μας, τους ε, μας από το πάνελ να απαντήσουν. Για πέντε λεπτά ο καθένας, εάν μπορείτε. Εάν θέλετε να πείτε πολλά, έχετε και απλώς τις ερωτήσεις, αλλά στην ουσία έχετε πέντε λεπτά ο καθένας. Η κυρία Βόλτσουκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις συναρπαστικές ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Νομίζω να ξεκινήσω από την ευρύτερη εικόνα, την οποία δεν είχα χρόνο να την ε, σχεδραφίσω. Αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει τώρα είναι η κατάρρευση της ε, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, μέρος δεύτερο. Η Ουκρανία έχει γίνει το, η σκηνή, το παλικοσένικο που αυτό εκτιλήσεται. Και αλλάζει και η σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Βλέπουμε παλιότερα στοιχεία της έννοιας του κράτους και του έθνους που ήταν καθοριστικά στην κατάρρευση της ε, Σοβιετικής Ένωσης να ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια μας. Βλέπουμε τις περιοχές που θέλουν να απομακρυνθούν. Έχουμε τρεις χώρες στην ουσία οι οποίες έχουν υπογράψει συμφωνίες σύνδεσης που όμως έχουν τάσεις αποσχιστικές εντός της επικράτειάς μας, της επικράτειάς τους. Βλέπουμε λοιπόν την Ρωσία να είναι παρούσα και με τις πυρηνικές ε, εξελίξεις έχουν ε, πια εξαλειφθεί όλες οι ψευδεστήσεις για την επικράτηση στον προεσοβιετικό χώρο. Αυτό ήταν ίσως το μεγαλύτερο κακό που μπόρεσε να κάνει η Ρωσία κατά των δικών της των συμφερόντων. Ήμουν στην Αρμενία πριν από δύο εβδομάδες και πραγματικά έμεινα έκπληκτη, γιατί παρά το γεγονός ότι πέντε μήνες μετά την απόφαση του Αρμένιου Προέδρου ο καθένας σε κάθε αρμενικό υπουργείο μιλούσαν περισσότερο για την ε, συνεργασία με, την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά με, την, με τις χώρες της Ευρασιατικής Θελωνιακής Ένωσης. Και στην Αρμενία δεν ήθελαν ούτε καν να ξέρουν λεπτομέρειες περί σύνδεσης. Αυτό δείχνει πώς η έλξη μπορεί να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και ότι χρειάζεται να σκεφτούμε πάρα πολύ, να μελετήσουμε το πρόβλημα για να δούμε πού ακριβώς ε, τι θέση παίρνει η Ρωσία σε σχέση με τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας. Είναι διαφορετικό το γεωπολιτικό και το στρατηγικό ε, τοπίο σήμερα. Πρέπει να συντονίσουμε τις ενεργειές μας ιδίως ως προς και στην ενδιάμεση ε, συμφωνία της σφαιρικής και βαθιάς συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών. Οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών έχουν να κάνουν με την προσέγγιση ε, προς το κοινωτικό κεκτημένο. Κατά 89% είχαμε ε, να υπάρχει στην Ουκρανία, αλλά όχι η ανάλυση κόστου ωφελίας για τις χώρες της Βαλτικής. Όμως, κυρίως ένας κατάλογος προτεραιοτήτων και το τι μεταρρυθμιστικά μέτρα χρειάζονται ώστε οι αναλύσεις κόστου ωφελίας για τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας μπορεί να πάρουν σάρκα και οστά και μάλιστα σύντομα και όχι στο μακροπρόθεσμο μέλλον. Ξέρουμε από όλε τι μελέτε ότι οι συμφωνίε τη Ανατολική Γειτονία θα επιτρέπουν την ανάπτυξη και είναι ωφέλιμε για τι χώρε. Αλλά υπάρχει ένα βραχυπρόθεσμο κόστο. Και αντί να έχουμε συγκεκριμένα εργαλεία για να αναχαιτήσουμε το κόστος αυτός με συγκεκριμένη αλληλουχία και ε, ιεράρχηση αναγκών ε, δεν προσφέρουμε κάτι, γιατί οι Ουκρανοί και οι Μολδαβοί παραγωγοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό. 50% του κόστους ε, της ε, πρόσληψης του κοινοτικού κεκτημένου είναι, είναι κάτι που πρέπει να το αναλάβουν οι επιχειρήσει των χωρών αυτών. Ε, αυτό λοιπόν ισχύει και στην Ουκρανία. Και να επικεντρωθώ ίσως στην Ανατολική και Νότια Ουκρανία. Πού θα σταματήσει η Ρωσία. Ίσως ούτε καν εκεί. Υπάρχει και ένα εφιαλτικό σενάριο που ελπίζω να μην υλοποιηθεί. Όμως βλέπουμε και πραγματικά βασίζομαι και στο κέντρο των ευρωπαϊκών και ρωσικών μελετών, στους συναδέλφους και τις γνώσεις τους και έχω ακούσει και από άλλους ειδικού περί Ρωσίας, ότι το σενάριο αυτό προγραμματίζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ότι σε πολύ συμπυκνωμένο χρονικό διάστημα έχει γίνει η σύλληψή του, αλλά η προώθηση της Ρωσίας ε, στην περιοχή αυτή δεν είναι κάτι το καινούριο. Είναι κάτι που δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία. Το βλέπουμε να συμβαίνει στην Ανατολική και Νότια Ουκρανία. Οι περιοχές αυτές με αποσχεστικές τάσεις είναι κάτι που βλέπουμε να ε, συμβαίνει στην πράξη, στην υπερνηστερία, στην Νότια Ουκρανία. Υπάρχει μια τάση της αναβίωσης της ε, Ρωσικής Συνομοσπονδίας με πρόσβαση μέσω της ζώνης, γεωγραφικής ζώνης αυτής από την Νότια Ουκρανία και την Υπερπιστηρία προς τις Αυτά δεν είναι αναγκαίο ότι θα συμβούν κατά αυτόν τον τρόπο και δεν έχουν να κάνουν μόνο με τους αγωγούς και την ε, οικοδόμηση αγωγών, αλλά ενδεχομένως και με την καταστροφή αγωγών και διάβλων η Ρωσία και αυτό είναι που με ανησυχεί είναι τι θα γίνει αν αυτοί οι αγωγοί ε, ανατιναχθούν και μπορέσει η Ρωσία να εισβάλλει κανονικά στην Ουκρανία. Αυτό λοιπόν που με θλίβει είναι ότι το BBC ε, στην αναμετάδοση της Ρωσίας έπαυσε να λειτουργεί στη Ρωσία. Βλέπουμε τι εικόνα αυτό μας δίνει για, τη δράση τους. Ευχαριστούμε κύριος Κάσιερ. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω ίσως με το τελευταίο ερώτημα για τα κατά πόσο αυτό το δημοψήφισμα ήταν φτημένο. Ε, Θα πρέπει να σκεφτούμε μακροπρόθεσμα την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και αυτή η κατάσταση πήρε καιρό να δημιουργηθεί. Το πώς τα εκλαμβάνουμε όλα αυτά έχει μεγάλη σημασία. Αυτή η αντιμελόπιτα, αυτή η αντιπαλότητα, αυτός ο ανταγωνισμός είναι κάτι που έτσι το αισθάνθηκε η ρωσική κυβέρνηση. Γι' αυτό έχει επιβάλλει αυτά τα μέτρα. Υπάρχει και μια διάσταση ενοχής, αλλά λύση δεν υπάρχει, πέρα από το να αναζητήσουμε λύσεις που όμως αυτές τις σημερινές συνθήκες φαίνεται να είναι απίθανες. Η οικοδόμηση λοιπόν εμπιστοσύνη είναι κάτι που θα πρέπει να το επιδιώξουμε σίγουρα στο μέλλον. Τι είδους ε, γείτονα θέλουμε, ένα μια τόσο μεγάλη χώρα όπως η Ρωσία, μια χώρα με ένα τόσο έντοξο παρελθόν που φοβάται να ταπεινωθεί, θα τις επιβάλλουμε εμείς τη δική μας αντίληψη για τα πράγματα, τι κυρώσεις θα επιβάλλουμε και τι κυρώσεις μπορεί να μας επιβάλλει η Ρωσία. Και από την άλλη είναι αναπόφευκτο να επιβληθούν τέτοιες κυρώσεις, Διότι έχουν ξεπεράσει κάποια όρια και αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε με, το σημερινό ευρωπαϊκό, με τα σημερινά ευρωπαϊκά δεδομένα. είναι, ήταν τόσα εκατομμύρια άνθρωποι σε συνθήκες επανάστασης ε, κατά ενός διαφθαρμένου καθεστώτος. Αυτό που με τον ένα τον άλλο τρόπο να ληφθεί υπόψη. Άρα η Ρωσία εκλαμβάνει τα γεγονότα αυτά σαν μια προσπάθεια αποδυνάμωσής της και μόνον. Οπότε τι μορφή συνεργασίας θα μπορούσαμε να προβλέψουμε. Δεν ξέρω αν ο ρεαλισμός είναι πιο, το, το μεγαλύτερο, το πιο σημαντικό ε, ρεύμα σκέψης ε, παγκοσμίω, όμω σίγουρα χρειάζεται οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Σχέσεων εμπιστοσύνη για να ξεπεραστεί αυτό το κλίμα. Αν αυτό θα γίνει με τον Πούτιν δεν είμαι βεβαίω, δεν είμαι πολύ αισιόδοξο, όμω πρέπει να σκεφτούμε και την υπόλοιπη Ρωσία εκτό από εκείνον. Και είμαι πεπισμένο, για να αναφερθώ και στι υπόλοιπε ερωτήσει, ότι η πολιτική του Πούτιν μπορεί να γίνει μπούμεραγκ η Ρωσία είναι πολύ πιο αδύναμη από το ρόλο που προσπαθεί να διαδραματίσει και αυτό φαίνεται εν τέλει και οικονομικά είναι ακόμη πολύ ευάλωτη. Είδαμε τι πτώση υπήρχε τουλάχιστον ε, κατά 25% από την αρχή της κρίσης και μπορεί και τα πράγματα να αλλάξουν λόγω της πίεσης των, ε, της κοινότητας των επιχειρηματιών εντός Ρωσίας. Μπορεί λοιπόν η Ρωσία να πληγώσει πολύ περισσότερο τον εαυτό της από ό,τι προσπαθεί να πλήξει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, για την Ουκρανία. Ε, υπάρχει μια ολόκληρη προπαγάνδα από τη ρωσική πλευρά και σε αυτό βασίζεται με το κόμμα του Φερμόντα που είναι ε, από τα πιο ακραία και εξταμιστικά και συμμετέχει στην κυβέρνηση αυτό. Είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε και θα το δούμε μετά τις προεδρικές εκλογές. Αλλά θα, υπάρξει, θα υπάρξουν εκλογές και για τη Βουλή. Οπότε εκεί θα πρέπει να προκύψει μια κυβέρνηση νομιμοποιημένη από δημοκρατικές εκλογές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παράξενη κατάσταση. Ένα κοινοβούλιο, ακριβώς το ίδιο με την πλειοψηφία που στηρίζεται το Γιαννουκόβιτς. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε κατά πόσο αυτή η κατάσταση μπορεί να είναι σταθερή και, ε, και θετική για το δημοκρατικό μέλλον της Ουκρανίας. Θα πρέπει λοιπόν να λυθεί το κοινοβούλιο και να ε, προκηρυχθούν εκλογές. Ένα πρώτο βήμα για να δημιουργηθεί μια σωστή Ουκρανική κυβέρνηση. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ κύριε Σπιτιά. Με όλο το σεβασμό κύριε Πρόεδρε, αν υπήρχε μόνο ο ρεαλισμός και αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε, δεν είμαι σίγουρος αν θα είχε επανενωθεί η χώρα μου ή αν θα είχαμε πολλά νέα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και την αξία, τη βάση της αξίας, την αξία της δημοκρατίας του κράτους δικαίου. Αυτό έχει μεγάλη σχέση και θα ήθελα να το τονίσω ότι οι συμφωνίες σύνδεσης δεν είναι μόνο συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου, έχουν και μεγάλο υπόβαθρο στις αξίες στις οποίες βασιζόμαστε, ιδιαίτερα τα συνδετικά στοιχεία, αυτά που μας συνδέουν. Και αυτό ίσως να είναι ο πιο μεγάλος πόλος έλξης και όπως είπε και ο κύριος Καζίρ, εκατοντάδες χιλιάδες ε, Ουκρανοί έχουν ξεχυθεί στον δρόμο όχι επειδή αγαπούν τόσο πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επειδή θέλουν να βγουν από μια μεταβατική κοινωνία που χαρακτηρίζεται από διαφθορά, όφελος ε, από τους νόμους για τους λίγους και τυχερούς προτιμούν ένα κράτος που θα ωφελεί τους πολίτες και αυτό είναι η ουσία. Και αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, ας είμαστε ρεαλιστές. Ας δούμε ότι υπάρχει παγκοσμιοποίηση, ότι θα πρέπει να είμαστε ικανοί και ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι να είμαστε, να φοράμε παροπίδες και να περιοριζόμαστε στον περιφερειακό ανταγωνισμό. Αυτό είναι σημαντικό τόσο για τη Ρωσία αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει περισσότερο και πιο στενά να συνεργαστούμε για την νεολαία και για τους πολίτες όλους είναι έντονη αυτή η διασύνδεση. Γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η διάσταση. Δεν είναι θύματα της προπαγάνδας της τηλεόρασης. Ξέρουμε ότι είναι παγκόσμια η κοινωνία. Για κάποια σχόλια των Ευρωβουλευτών. Καταρχάς, δεν αφορά την κυρία Κουψέβα. Μιλήσατε για την επιρροή των εξτρεμιστικών κομμάτων. Θα ήθελα να τονίσω στο σημείο αυτό ότι η κυβέρνηση εκλέχθηκε με 371 μία ψήφους συνταγματική πλειοψηφία, το οποίο περιλαμβάνει και πολλά κόμματα των, του, του κόμματος των περιφερειών, το οποίο θεωρήθηκε ότι θα είχε πιο καλές πιθανότητες ε, στις μελλοντικέ εκλογές αν δεν συμμετείχε στην κυβέρνηση. Να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί, να μην θεωρήσουμε ότι είναι κατά οποιονδήποτε τρόπο ε, μη νόμιμη η κυβέρνηση αυτή. Έγιναν ε, προεδρικές εκλογές και κοινοβουλευτικές εκλογές προσφάτως. Κύριε Τάνοκ ρωτήσατε κατά πόσον έχουν επιβληθεί σωστέ κυρώσει. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπα και προηγουμένως. Η απάντηση και η προσέγγιση των αρχηγών κυβερνήσεων και των Υπουργών Εξωτερικών είναι ότι πρόκειται για την έναρξη των κυρώσεων. Κυρώσεων που μπορεί να κλιμακωθούν. Δεν θέλουμε να μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο, αλλά θέλουμε να δώσουμε ένα σαφές και χειρό μήνυμα προς την Ρωσία. Έχει οριστεί και μια τρίτη φάση που από αρχηγού κυβερνήσεων και κρατών όταν μιλούν για επιβολή κυρώσεων οικονομικών και μη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των, της Ρωσίας. Κατά πόσον είναι ε, ενιαίος ο αντίκτυπος στην ε, Ρωσία. Υποθέτω ότι η, ο αποσταθεροποιητικός παράγοντας είναι αρκετά σημαντικός. αν θεωρηθεί ότι η Κρυμαία έχει φύγει από την Ουκρανία, αυτό μόνο να ενδυναμώσει μπορεί τις προδοτικές και τις δυνάμεις που υποστηρίζουν τη Δύση και την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία. Είπατε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι πιο άκαμπτες και αυστηρές. Είναι πιο εύκολο να το κάνουν όμως, γιατί έχουν πολύ πιο περιορισμένες οικονομικές σχέσεις και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία. Άρα ως εκ τούτου, είναι πολύ πιο διαφοροποιημένη η προσέγγιση μας. Το πολιτικό μήνυμα, ωστόσο, είναι ακριβώς το ίδιο σε ό,τι αφορά την παραβίαση της επικυριαρχίας και της εδαφικής αικαιρεότητας της Ουκρανίας. Ο η κυρία Κρόνμπεργκ είπε ότι θα πρέπει να είμαστε πιο προετοιμασμένοι για το μέλλον και να δούμε πώς αντιλαμβάνεται η Ρωσία τις πολιτικές μας. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Το είπε και η κ. Καζιέ. Παρά το γεγονός ότι είμαστε πεπισμένοι για το ότι είναι δίκαιες οι πολιτικές μας, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους Ρώσους ομολόγους μας, γιατί θεωρούν ότι οι πολιτικές μας είναι στραμμένες κατά της Ρωσίας. Πεπισμένοι ότι και από οικονομικής αλλά και πολιτικής άποψης αυτό θα μας ωφελήσει αμφότερους. Είναι δυναμική όμως αυτή η προσέγγιση και είναι ισχυρή η πεποίθησή μας και η πίστη μας στην, ε, στον ιδιωτικό τομέα. Από την άλλη υπάρχει και μια στατική προσέγγιση, δεσμεύσεις και υποσχέσεις του παρελθόντος, κατηγορίες από το παρελθόν, αλλά αυτό είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί μόνο να βλάψει και όχι να ωφελήσει. Ο κ. Βιλιάνσε έθεσε ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα κατά πόσο οι πολίτες της Ουκρανίας θα ωφελούνταν από την απελευθέρωση των θεωρήσεων αν ζουν στην Κρυμαία. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι σαφές ότι αν δίναμε τέτοια απελευθέρωση από το καθεστώς των θεωρήσεων, ο οποιοδήποτε πολίτης της Μολδαβίας θα μπορούσε να υποφεληθεί από την απελευθέρωση των θεωρήσεων με τη χρήση του διαβατηρίου του. Το ίδιο θα σήμαινε και με τους Ουκρανούς πολίτες από τη στιγμή που θα είχε τέτοιο διαβατήριο. Και αυτό φυσικά δεν εξαρτάται από τη γλώσσα που θα χρησιμοποιούσε το άτομο αυτό. Αυτό ως απάντηση στις ερωτήσεις που τέθηκαν. Σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να τονίσω ότι ο πολιτικός ρεαλισμός έχει να κάνει με εξουσία, με την εξουσία. Η εξουσία ασκείται είτε μέσω α, ομάδων είτε μέσω προσέγγισης και προσέλκυσης. Αλλά παράλληλα πώς μπορούμε να επωφεληθούμε α, από, τις, ε, από την πολιτική της προσέλκυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν από την άλλη πλευρά έχουμε τα τάγκς. Και η δικιά μας ε, λογική για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και εδώ οι γεωπολιτικές σκέψεις έχουν, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο. Όχι μόνο οι ευρωπαϊκές αξίες, αλλά και αυτές οι περιστάσεις. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν. Ο κύριος Μπάλας έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ. Έχουν ήδη απαντηθεί περισσότερες ερωτήσεις. Εγώ θα ξεκινήσω με αυτά που είπατε εσείς κύριε Πρόεδρε, ότι εδώ έχουμε την ήπια δύναμη απέναντι στην σκληρή δύναμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί την ήπια δύναμη, soft power. Και επειδή κνεί όχι μόνο οικονομικό ρεαλισμό, αλλά θέλει να γίνει δελεστικό μοντέλο, θελκτικό μοντέλο και από οικονομική και από κοινωνική άποψη μοντέλο και παράδειγμα προς για οποιαδήποτε χώρα θα ήθελε να την μυθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεται πολιτικές τύπου Ρωσίας, τουλάχιστον αυτής που χρησιμοποιήσει η Ρωσία το τελευταίο καιρό για να προσελκύσει μέλη στην Τελωνιακή Ένωση. εμείς έχουμε πρόβλημα να, μην δημιουργούμε φρούδες ελπίδες ε, για προσχώρηση στις ε, χώρες με τις οποίες έχουμε συνεργασία. Περισσότερο αυτό ήταν ένα θέμα για μας. Επίσης, ε, μια και μιλούμε για οικονομικά μοντέλα, θέλουμε να δημιουργήσουμε ελπίδες για τις χώρες που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το εξυγχρονιστικό δικό μας οικονομικό μοντέλο και ελπίζω ότι θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Αυτό έγινε στις αναδυόμενες οικονομίες. αν δείτε τι συνέβη στην ρωσική οικονομία, δεν μπορείτε πια να τη χαρακτηρίζετε ως αναδυόμενη οικονομία ή δυναμικά αναπτυσσόμενη οικονομία. Και αυτό είναι αρκετά αρνητικό ήδη για τους ίδιους τους Ρώσους, αλλά επίσης και για τους υπόλοιπους εταίρους ε, ε, της Ανατολής. Και Γι' αυτό ενδιαφέρονται και για όλο και πιο στενές σχέσεις με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά αυτά που είπε η κυρία Λιούπτσεβα για τα λάθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την δημιουργία των σχέσεων ανατολικής εταιρικής σχέσης ε, και τα λάθη που κάναμε απέναντι στη Ρωσία. Όπως είπα και προηγουμένως, εμείς ε, ήμασταν ανοιχτοί για συζήτηση με τη Ρωσία, αλλά δεν έδειξε αντίστοιχο ενδιαφέρον η Ρωσία για συζητήσεις μαζί μα. Ενώ η Ρωσία ενδιαφέρθηκε περισσότερο για τριμερείς διαλόγους. Τριμερείς διαλόγους ε, από την άποψη ότι να έχουμε Ουκρανία, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία. Εμεί δεν συμφωνούμε. Δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι ο σωστό τρόπο σύντηση μεταξύ κυρίαρχων χωρών. Δεν θεωρούμε ότι η Ουκρανία είναι μια χώρα που χρειάζεται το μεγάλο αδελφό για να την προστατεύσει ή ε, άλλε χώρε που θα είναι προστατευτικέ απέναντι τη. Εμεί θέλουμε διμερεί σχέσει με την Ουκρανία και είμαστε έτοιμοι για τέτοιε διαπραγματεύσει. και είμαστε έτοιμοι για διάλογο με τη Ρωσία, θεωρεί ότι της, αλλά σίγουρα δεν, θα, δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ιδιαίτερα δικαιώματα της Ρωσίας απέναντι ε, σε χώρες ε, που αποκαλεί κάπως πατερναλιστικά τους ε, κοντινούς της γείτονες. Τώρα, με δεδομένες τις παρούσες δυσκολίες, τι θα κάνουμε με τις τρεις κυριότερες χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Τώρα, ως προς την Ουκρανία, όπως είπαμε, υιοθετήθηκαν ε, μέσα για μονομερή εφαρμογή της, ελευθε... της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών κατά πάσα πιθανότητα τις επόμενες εβδομάδες, αν καταφέρουμε να τηρήσουμε αυτό το στενό χρονοδιάγραμμα για να τεθεί σε ισχύ ολόκληρη η συμφωνία, ώστε να ανοίξουμε την ε, ενιαία αγορά, την ευρωπαϊκή αγορά προς την Ουκρανία. Αυτό έχει ήδη αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ήδη έχουμε και την κανονιστική εναρμόνιση και δεν συμφωνώ με εκείνους που είπαν ότι είναι ένα ουτοπικό και υπερβολικό βάρος, άχθος. Τα ευρωπαϊκά προϊόντα, μάλλον ε, τα προϊόντα τρίτο χώρο θα πρέπει να πληρούν τι δικέ μα υψηλέ προδιαγραφέ υγειονομικέ και άλλε. Αλλιώ δεν μπορούν να, να εισέλθουν στον ε, νέο χώρο. Επίση, προσφέρουμε τεχνική αρρωγή στι χώρε αυτέ για να μπορέσουν να εκπληρώσουν αυτέ τι προδιαγραφέ και να χρησιμοποιήσουν τι ε, δασμολογικέ προτιμήσει που χορηγούμε ω Ευρωπαϊκή Ένωση και να διευκολύνουμε αυτέ τι χώρε να ε, προσχωρήσουν. Επίση, παρόμοια μονομερή μέτρα εφαρμόσαμε και για τη Μολδαβία. που έχει αυτόνομες εμπορικές ε, προτιμήσεις. Και επίσης και η Γεωργία είναι η τρίτη χώρα που απολαμβάνει μονομερείς προτιμήσεις με βάση το καθεστώς γενικευμένων ε, δασμολογικών προτιμήσεων ΣΥΝ. Έχει ειδικέ δασμολογικές προτιμήσεις δηλαδή για χώρες όπως η Μολδαβία που μπορούν ε, μόνο μερός να ανοίξουν την αγορά τους. Ευχαριστώ. Αυτό είναι ενδεικτικό της ελαστικότητας που επιδεικνύουμε και που χρειάζεται και τώρα αν θέλουμε να προσαρμόσουμε τους μηχανισμούς μας και, τα εργαλεία μας σε καταστάσεις που διαμορφώθηκαν στην πορεία. Πάντως χαίρομαι για την ευκαιρία που έχουμε για ανταλλαγή, για την ευκαιρία που είχαμε για ανταλλαγή απόψεων και για τη δημόσια κράση και θα δώσω το λόγο τώρα στον συνάδελφο από την ε, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου για να αντλήσει κάποια συμπεράσματα. Καταλήξαμε σε πολλά συμπεράσματα σήμερα, αλλά ένα είναι σίγουρο. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε, να φροντίσουμε μάλλον να μην δώσουμε κατόπιν εορτής και εκ των υστέρων τις προτάσεις και τις συστάσεις μας. Γιατί αυτό που συνέβη στην Ουκρανία και στην Κρυμαία δείχνει ότι θα πρέπει να είμαστε διορατικοί και να προβλέπουμε μερικά πράγματα ε, και όχι όταν η Ρωσία μας φέρνει την πρώτη γεγονότων και να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις να επαναληφθούν στο μέλλον. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω. Σας ευχαριστώ θερμά λοιπόν. Συνάδελφοι, παρακαλώ. Όσους δεν συμμετέχουν στις περαιτέρω εργασίες της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων να εγκαταλείψουν αθόρυβα την αίθουσα γιατί έχουμε αρκετά σημεία στην ημερήσια διάταξή μας και θα πρέπει να τα διεκπαιρεώσουμε όλα. Περνάμε τώρα στο σημείο 5 της της διάταξης, τις συστάσεις προς το Συμβούλιο σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας. Δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Πέτερλε. Παρακαλώ κύριε εισηγητά. Eh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερος επειδή έχουμε φτάσει πια σε μια τέτοια χρονική στιγμή όπου η στάση μας εναντί αυτής της συμφωνίας έχει αποσαφινιστεί. Ευχαριστώ τους ε, σκιώδεις που ε, ήταν διαλλακτικοί και μπορέσαμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις. Νομίζω ε, τα στοιχεία που προέκυψαν στο μεταξύ συνάδουν με το γενικότερο πνεύμα της έκθεσης και ελπίζω τα περισσότερα να γίνουν δεκτά και από τους συναδέλφους. Εγώ δέχτηκα τις τροπολογίες που αποσαφηνίζουν, ενδυναμώνουν την έκθεση, ώστε να δοθούν κάποιες σαφείς συστάσεις προς τους διαπραγματευτές. Κατα... Τοποθετήθηκαν ειδικά ως προς τις τροπολογίες που κάνουν την έκθεση ε, ε, υπερβολικά ε, λεπτομερή σε σχέση με κάποια πράγματα που μπορεί να συμβούν. το θέμα δεν είναι κατά πόσον θα επηρεάσουμε τις τελικές αποφάσεις, αλλά κατά πόσον η διαπραγματευτική εντολή ε, μπορεί να φέρει τις ε, αλλαγές που επιθυμούμε. Η συνεργασία εδώ είναι καθοριστική σημασία και η έκθεση αυτή τονίζει τις ε, φιλοδοξίες μας και τις επιθυμίες μας για μια τέτοια περιοχή, ανοίγοντας και νέες δυνατότητες συνεργασίας όπως φαίνεται από τις τροπολογίες που αποβλήθηκαν. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που υπήρξε και μια σημαντική δήλωση από τον Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας για την συνέχιση των σχέσεών μας και για κάποιο ζήτημα που αυτή τη στιγμή μας έχει δημιουργήσει προβλήματα. Ένα, μια δήλωση που έγινε δεκτή με μεγάλη ανακούφιση και από την Νότια Κορέα. Οπότε η συμφωνία αυτή που βλέπουμε έχει θετική επίδραση και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Δεν χρειάζεται λοιπόν να περάσουμε σε προφορική τροπολογία για τον ιστορικό ρεβιζιονισμό. Ε, τώρα για τις τροπολογίες η πρώτη είναι μια πολιτική ε, διευκρίνηση. Νομίζω δεν χρειάζονται περισσότερο, ε, περισσότερες διευκρινήσεις για το ζήτημα της διασύνδεσης. Οι διπλωματευτές θα αναζητήσουν την καταλληλότερη διατύπωση μια διατύπωση που θα μπορεί να είναι αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. ώστε να υπάρχει κατάλληλη ε, διασύνδεση. Ε, αυτά λίγο πολύ, Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω για αυτή την εισαγωγική μου παρέμβαση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Βρίσκομαι σε μια περίεργη θέση, γιατί είμαι και σκιώδης εισηγητής και από τη δική μου ομάδα δεν υπάρχει κανείς άλλος στην αίθουσα. Θα πρέπει λοιπόν να το αντέξετε. Πρέπει να μιλήσω και με αυτή μου την ιδιότητα και να πω ότι μέρος του προβλήματος σε αυτό το τομέα, όπως τα ξέρετε, είναι ότι όλα τα μέρη προσπαθούν να επανερμηνεύσουν το παρελθόν. Και όπως θα γνωρίζετε, ε, κοιτάζοντας προς το μέλλον, θα πρέπει να έχουμε και μια τοποθετήση σε σχέση με το πραγματικό θα κλείσω τώρα με αυτά και θα ήθελα να, να δώσω το λόγο στον κύριο Μπουτικόφερ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή μα, τον κύριο Πέτερλε. Όντω, είχαμε συζητήσει όπου προσπάθησε ο κύριος Πέτερλε προσπάθησε να καλύψει τις ιδέες και τις απόψεις που εκφράστηκαν από δική μας πλευράς. Ε, μπορέσαμε συστηματικά να συμβαζόμαστε. Γι' αυτό ήθελα να τονίσω μόνο μερικά σημεία τα οποία ε, έχουν απασχολήσει ειδικώ εμάς. Το πρώτο αφορά την πρώτη τροπολογία η οποία αγγίζει το θέμα που αναφέραμε. Έχει αλλάξει η κατάσταση σε σχέση με αυτό που μας απασχολούσε όμως με τις παλακίδες διότι ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός αποσχέθηκε να το διερευνήσει. Δεν είμαι βέβαια έτοιμος αυτή τη στιγμή να πω ότι έχω καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα. Παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα είναι τόσο ευαίσθητο που θα ήταν σημαντικό να μην παραλείψει το Κοινοβούλιο να το εντοπίσει. Τώρα για την πέμπτη τροπολογία ελπίζω ότι θα υπάρξει στήριξη για την ιδέα να διευρύνουμε το πεδίο συνεργασίας μας πέραν της ειρηνικής χρήσης πυρηνικής ενέργειας και μόνον όπως αναφέρεται. Η συγκεκριμένη πρόταση και φράση στα πλαίσια των συγκεκριμένων σχέσεων ίσως να ε, γίνει αντιληπτή ως μονομερής τοποθέτηση. Προσπαθούμε λοιπόν, θα πρέπει να προσπαθήσουμε εκεί λίγο να μεταβάλουμε το πεδίο. Με συγχωρείτε. Για την Τροπολογία 30. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αποσχολήσει αμφότερες τις πλευρές. Μια σφαιρική και συνολική απόκριση στις κλιματικές αλλαγές. Εδώ θα καλέσω τους συναδέλφους να συμφωνήσουν και με αυτήν την προσθήκη. Να αναφέρω τώρα ε, λίγα λόγια ακόμα για την προφορική τροπολογία επαριθμών 2 με συγχωρείτε, την πρώτη προφορική τροπολογία που αφορά την 2, την 4 που αφορά την 19 και την 10 που αφορά την 35, προσπαθήσαμε να προσαρμόσουμε την αρχική διατύπωση ώστε να φανεί ώστε να είναι και πιο εφικτό για τους υπόλοιπους συναδέλφους να ακολουθήσουν αυτή τη λύση. Ευχαριστούμε κύριο Πέτρελε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν ανέφερα τις συγκεκριμένες τροπολογίες που αποτέχθη η συμφωνία και για τη Φουκουσίμα και για άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την πυρηνική ενέργεια. Μιλούμε για την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικού σκοπούς. Ελπίζω ότι η συμφωνία θα επιτευχθεί και στην τροπολογία που υπάρχουν ακόμη κάποιες διαφωνίες και λόγω των νέων ε, γεγονότων που προέκυψαν. Ο κύριος Αλαφράγκα θέλει να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ. Λακωνικά κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να στηρίξω το έργο του κυρίου Πέτερλε και να συγχαρώ τον εισηγητή η έκθεση αυτή φυσικά θα πρέπει να ταινίζει το μέλλον και επειδή η Ιαπωνία είναι πολύ θετικός και επικοδομητικός εταίρος Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να βρούμε τρόπους για να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας. Μάλιστα, επειδή έχουμε και άλλους εταίρους και με την Ανατολική Γειτονία και με άλλες σημαντικούς παγκοσμίους εταίρους ε, όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία. Έχουμε εκκρεμίσει διαπραγματεύσει με το Μερκοσούρ. Κατοχυρωνόμαστε ως ε, παγκόσμιο εταίρο, οπότε θα πρέπει με τις καλύτερες δυνατές προποθέσει ε, να διεκπαιρεώσουμε, να κλείσουμε αυτή τη συμφωνία με την Ιαπωνία προς το αμοιβαίο συμφέρον και των δύο συμβολωμένων μέρων. Επίσης, στη συμφωνία μας θα πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην, στη ρήτρα της δημοκρατίας, στη δημοκρατική ρήτρα, γιατί αντικατοπτρίζει την προσήλωσή μας στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και όπως είπε ο εισηγητής θα πρέπει να καταφέρουμε να βρούμε μια διατύπωση που θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο, φυσικά μένοντας πιστοί ε, στις, ε, στους όρους και την παράδοση που ισχύει για τις διάφορες συμφωνίες. Πιστεύω ότι θα βρούμε το δρόμο, θα ξεπεράσουμε το εμπόδιο αυτό και επαναλαμβάνω την ε, υποστήριξη της πολιτικής μου ομάδας προς τον εισηγητή, τον κύριο Πέτρελε για την εξαιρετική του δουλειά και ευελπιστούμε ότι η έκθεση θα συγκεντρώσει μεγάλη πλειοψηφία στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της της διάταξης, σύσταση προς το Συμβούλιο για την 69η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Θα δώσω το λόγο στον κυρία Νέιτς που αντικαθιστά τον κύριο Λάμστορφ ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα στη συνεδρίαση. Δίνω λοιπόν το λόγο στην κυρία Νέιτς. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Αλεξάνδρ Λάμπστορφ συνέταξε τη σύσταση και το ψήφισμα και είχε συνομιλίες με τους και ηγετές των πολιτικών ομάδων προκειμένου να καταλήξει συμφωνία επί των συμβαστικών τροπολογιών. Έχουν μοιραστεί όλες αυτές οι προτάσεις, οι συμβαστικές. Οπότε είστε όλοι κατατοπισμένοι. Περιμένω τώρα τη, τον σχολιασμό αυτών των προτάσεων, τις αντιδράσεις σας και να επιστήσω την προσοχή σας το γεγονός ότι υπάρχουν και δύο ή τρεις προφορικές τροπολογίες που θα καταθέσει ο συγγετής ο κύριος Λάμστορφ. Η μία προφορική τροπολογία αφορά την τροπολογία 15 του κυρίου Σόλτς, προκειμένου να αντικατασταθεί ε, το female από το women, εκεί που λέμε θηλυκά, ε, από γυναίκες. Είναι πιο κομψή, κομψός όρος. Και επίση μια άλλη προφορική τροπολογία θα κατατεθεί για την τροπολογία 22 με πρόταση να τροποποιηθεί ένα τμήμα της τροπολογίας ε, από το αρχικό ε, κείμενο για το σημείο α που θα προβλέπει το εξής. Το σημείο α λοιπόν να συμβάλλει ε, παρακολούθηση και εφαρμογή της δήλωσης ε, της ε, συνάντησης υψηλού επίπεδου για το κράτος δικαίου της 24 Σεπτεμβρίου 2012 και να δει σε ποιο βαθμό μπορεί το κράτος δικαίου να συνδυαστεί με τις συνεχείς συζητήσεις και σκέψεις για τις αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας μετά το 2015. Αυτά προβλέπει το α. Ουσιαστικά επαναρχόμαστε στο αρχικό σημείο α. Επίσης ε, για την 51 του κυρίου Στίερ ε, προτείνουμε να συμπεριληφθεί ως προσθήκη στο Q, το αρχικό Q. Και επίσης ε, προτείνονται κάποιες αλλαγές στην τροπολογία 64 της κυρίας Μονής. Περιμένω τα σχόλια των συναδέλφων. Αν δεν υπάρχουν, το κείμενο θα ψηφιστεί με τη μορφή που έχει λάβει μετά τις συμβαστικές τροπολογίες και τη συμπερίληψη των προφορικών και άλλων τροπολογιών που δεν καλύπτονται από τις συμβαστικές. Ευχαριστώ κύριο Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την κυρία Νέιτς που αναπλήρωσε τον εισηγητή τον κύριο Λάμστορφ. Και εγώ εκπροσωπώ εδώ τον κύριο Πρέντα που είναι ο σκιώδης του ΕΛΚ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λάμστφορτ για την ε, αγαστή συνεργασία που είχαμε, για τη σύνταξη της, ε, του σχεδίου σύστασης και το συνεργάσιμο και διαλλακτικό του πνεύμα στη διάρκεια των συζητήσεων. Ο σκιώδης ηγητή ο κ. Πρέντα θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη συνένεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων προκειμένου να καθοριστούν οι προτεραιότητες μας εν ώψη της 69ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και τις προτεραιότητε μας, τις προτεραιότητες μας αυτές θα τις περιλάβουμε σε μία σαφή σύσταση που θα περιγράφει τα σημεία που μας ενδιαφέρουν. Ο κύριος Πρέντα μου ζήτησε να μεταφέρω τις παρατηρήσεις του για συγκεκριμένα σημεία. Κατά τη γνώμη του, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή των συστάσεων που, που έχουν ε, υιοθετηθεί στη συναντήση ψηλού επίπεδου για το κράτος δικαίου. Σε ό,τι αφορά την ειρήνη και την ασφάλεια, ο κύριος Πρέντα θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσουν οι περιφερειακές οργανώσεις ε, ε, ιδιαίτερα για την κρίση, όπως έδειξαν οι κρίσει στο Μαλί και στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ο ρόλο λοιπόν των περιφερειακών οργανώσεων για την υλοποίηση αυτών των στόχων και επίση ε, να υπογραμμίσουμε τη σημασία που έχει πρόληψη στα πλαίσια τη ευθύνη προστασία. Σε ό,τι αφορά τη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση με τα Ηνωμένα Έθνη, ο σκιώδη μα ηγητή επιμένει στην ανάγκη και μέσω και μακροπρόθεσμα ε, να επιδιώξουμε σε ένα νεωμένο ε, Συμβούλιο Ασφαλείας την όχι μόνο την δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μιλάμε ενιαία φωνή, αλλά και να έχουν έχει έδρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οντότητα σε ένα διευρυμένο Συμβούλιο Ασφαλείας. Γι' αυτό και ζητούμε να συμπεριληφθεί η τροπολογία 57 του κ. Μιγιάν Μον. Σε ό,τι αφορά τη... την εξέλιξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας μετά το 2015, ο κ. Πρέντα τονίζει την ανάγκη να έχουμε ένα ενιαίο και ευρύ πλαίσιο για την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας μετά το 2015 με σαφή κριτήρια εφαρμογής, συμπεριλαμβάνοντας ε, τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε θέματα ανάπτυξης και αηφορίας. Ένα συγκεκριμένο σχόλιο αφορά τη χρηματοδότηση αυτού του θεματολογίου της ανάπτυξης ε, για μετά το 2015. Κατά τη γνώμη του κ. Πρέντα, η θέση που αναφέρεται στην παράγραφο π του ψηφίσματος ίσως δίνει την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απρόθυμη να δεσμευτεί οικονομικά. Ενώ στην ουσία τα συμπεράσματα του Δεκεμβρίου του 2013 δείχνουν την ε, προθυμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δεσμευτεί σε μια αναπτυξιακή προσπάθεια και σε ένα αναπτυξιακό θεματολόγιο. Αλλά δεν ισχύει αυτή η προθυμία. Οπότε θα ήθελε ο κύριος Πρέντα να ζητήσει από τον εισηγητή τον κύριο Λάμστορφ να δεχθεί την, έκθεση, την τροπολογία του υπαριθμού 49 που δείχνει ακριβώς τη δεδηλωμένη ε, βούληση του, Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να στηρίξει την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας για μετά το 2015. Θα πρέπει να πάρω το λόγο εξ ονόματο τη κυρία Μουνή, που είναι μου είναι σκιώδη συγγετρία για το θέμα αυτό και θα ήθελα να συνοψίσω αυτά τα στοιχεία που μου ανέφερε. Μία σειρά τροπολογιών εισήχθησαν εξ ονόματο τη ομάδα μα, κατατέθηκαν από την ομάδα μα, αλλά υπάρχει και υποστήριξη από πλευρά τη ομάδα μα για όλες τις τροπολογίες που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών, 43-48 για την κυρία Σχάκια και για την τροπολογία υπεριθμών 44. Πρακτικά θεωρούμε ότι τα δικαιώματα των γυναικών αποτελούν ε, βασική προτεραιότητα όλων των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων και η ομάδα υποστηρίζει όλες τις εργασίες σε ό,τι αφορά τον ορισμό διεθνώ του κλιματικών προσφύγων. Σε ό,τι αφορά την Συρία, η ομάδα μας υποστηρίζει την σύσταση ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Διερεύνησης ε, για τη διερεύνηση όλων των ε, παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι θα πρέπει να προσαχθούν οι υπέτοι. Άρα, θα ήθελα να ζητήσω να μας πει η κυρία Νέιτς αν θέλει να πάρει το λόγο για να συνοψίσει. κυρία Νέιτς, ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις που έκαναν σε ό,τι αφορά το σαφή αίτημα των σκιωδών, του σκιωδούς ε, κυρίου Πρέντα για την ε, ε, τροπολογία 49. Θα πρέπει να το ελέγξω και να ζητήσω από τον συντάκτη της νομοδότησης να μας πει ποια είναι η θέση της. Δεν μπορώ έτσι αυθόρμητα να αποφανθώ, αλλά θα ήθελα εκ νέου να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για, για την συμβολή τους και νομίζω ότι θα φανεί αυτό αύριο στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρος. Και τώρα ας περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ξέρετε ότι αυτό θα ήταν η σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του Ιράν. Επειδή όμως ο συνάδελφος μου, η συνάδελφός μου Μαρία δεν είναι εδώ. Θα αναγκαστούμε λοιπόν να το αναβάλουμε το θέμα αυτό. Θα ψηφίσουμε χωρίς συζήτηση. Μια και δεν είναι εδώ πέρα η συγγήτρια. Η κυρία Σκάκα. Είστε σκιώδης. Πρόεδρε, πρόεδρε, είναι ένα θέμα αυτό. Ο κύριος Αλαφράγκα είναι πρώτος ή εσείς. Η κυρία Σκάκη, η κυρια σχακε Σκάκη. σχακε επι της διαδικασίας επιτρέψτε μου θα μπορούσαμε να το κοινοποιούμε λίγο πιο νωρίς αν ε, πρόκειται να απουσιάσουν οι συγητές. Γιατί ένας λόγος που βρίσκομαι εδώ στην αίθουσα είναι η σύσταση ακριβώς για το Ιράν. Και είναι φυσικά σημαντικό το θέμα αυτό. Καταλαβαίνω ότι οι συνάδελφοι μπορεί να έχουν άλλες υποχρεώσεις, αλλά είναι θέμα τουλάχιστον συνολικότητας να το ανακοινώνουν αυτό εγκαίρως. Έχετε δίκιο, λέει ο πρόεδρος, αλλά δυστυχώς έτσι έχει η κατάσταση. Πολιτικός ρεαλισμός ονομάζεται αυτό και πρέπει να το Ο κύριος Αλαφράγκα. Θα ήθελα να πω ότι η κυρία Σάκε έχει απόλυτο δίκιο και επίσης θα ήθελα να πω ότι δεν είναι κατά τη γνώμη μου σωστή διαδικασία να ετοιμάσουμε και να ψηφίσουμε αύριο χωρίς προηγούμενη συζήτηση. Δεν το δέχομαι. Ο σκιώδης ηγητής ε, της πολιτικής μου ομάδας ε, και εκείνος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί αλλά ανέθεσε σε μένα να τον εκπροσωπήσω. Το ίδιο κάνουν και άλλες πολιτικές ομάδες. Δεν είναι σωστό ούτε αρμόζουν να ψηφίζουμε χωρίς να έχει προηγηθεί συζήτηση. Εγώ θα έλεγα να το συζητήσουμε. Έστω και ερήμη της ηγητής. Λυπούμε για την απουσία της. Και Λυπούμε ακόμη περισσότερο που δεν ανέθεσε σε άλλον ε, ευρωβουλευτή να την αντικαταστήσει. Αν εσείς αποφασίσετε να μην γίνει συζήτηση, τότε και αύριο δεν επιτρέπεται να γίνει ψηφοφορία, γιατί αυτό προϋποθέτει μία απαράδεκτη τροποποίηση των κανόνων. Όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Σάκη, ε, κανονίσαμε το πρόγραμμά μας. Ε, όλοι αυτό κάναμε και άλλες πολιτικές ομάδες. Με βάση μια διαδικασία που έχει προκαθοριστεί και που περιλαμβάνεται στην ε, ημερήσια διάταξη. Δεν είναι αρμόσα μια τέτοια κατάσταση και διαδικασία. Ή θα συζητήσουμε σήμερα, ή αν δεν συζητήσουμε σήμερα, ούτε και αύριο μπορούμε να ψηφίσουμε. Δεν είναι δυνατόν να ψηφίζουμε χωρίς να έχει προηγηθεί συζήτηση που όμως είχε προγραμματιστεί. Από ό,τι ξέρω έγινε συνάντηση των σκιωδών εισηγητών για την ε, έκθεση αυτή και ξέρω ότι υπάρχει μια κάποια συμφωνία. Πολιτικός πώς λοιπόν έχουμε καλύψει κάποιο από το έδαφος. Μπορούμε να κάνουμε συζήτηση χωρίς την εισηγήτρια. Μπορείτε να παρουσιάσετε την θέση σας, το μπορεί να κάνει και η κυρία Σχάκε, αν επιμένετε. Και φυσικά θα διαβιβάσουμε τα στοιχεία που θα αναφέρεται στην εισηγήτρια. Και αυτό είναι ο μοναδικό τρόπο που μπορούμε να λύσουμε την ε, κατάσταση αυτή. Ή άλλω δεν θα μπορέσει να περάσει το θέμα αυτό στην ε, τρέχουσα θητεία. Και ξέρετε ότι δεν είναι η δική μα η ομάδα που καταρτίζει την έκθεση. Το, το θέμα το επιτάσσει. Το Ιράν. Καταλαβαίνετε. Ξέρετε ότι είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή των διαπραγματεύσεων. Και ξέρετε, νομίζω ότι αυτό είναι ο συμβιβασμό ε, εφόσον και αν τον αποδέχεστε. Κύριε Σαλαφράγκα. Κύριε Πρόεδρε, αυτό ακριβώ είπα και εγώ. Γιατί ξεκινούμε από τη βάση ότι συμμετέχουμε σε ένα δημοκρατικό όργανο, όπως είναι η Επιτροπή ΑΦΕΤ. Είναι θεμητό να έχει ανηλυμένη υποχρέωση η συγκήτρια είναι απασχολημένη κάπου αλλού, αλλά δεν δικαιολογείται η αναβολή, η ακύρωση της συζήτησης γιατί αν ε, είχαμε τέτοια διαδικασία σε όλες τις εκθέσεις, τότε δεν χρειάζεται καν να συνεδριάζουμε. Να αφήνουμε τους και και τον εισηγητή να τα συμφώνουν και εμείς περιτεύουμε. Πιστεύω ότι αν θέλετε να ψηφίσουμε αύριο, το μόνο που ε, επιτρέπεται, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε συζήτηση τώρα. Νομίζω ότι είναι μια πρόταση που πλησιάζει και με... είναι πανομοιότυπη με τη δική σας. Μάλιστα. Μάλιστα, λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση. Διαδικαστικό, μάλιστα. Ισκιώτης λοιπόν, πρώτη. Η κυρία Κρόμπερκ. Σκιώδης, η έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε και χαίρομαι που γίνεται αυτή η συζήτηση. Καταρχάς να καλωσορίσω και εγώ και η ομάδα μου την έκθεση είναι σε πολύ επίκαιρη χρονική στιγμή. Πάνε καλά οι διαπραγματεύσει. Μάλλον προχωράνε οι διαπραγματεύσει. Μόλι επισκέφθηκε η κυρία Άστον το Ιράν. Είναι σημαντικό. ότι δεν ε, τονίζεται στην έκθεση κάτι το οποίο ενδεχομένως να επιδεινώσει την ε, κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει να δώσουμε το περιθώριο να επιτευχθεί μια τελική συμφωνία να μην ζητάμε δηλαδή τελική και οριστική πάυση της εμπλουτισμού ουρανίου. Δύο τρία πράγματα θα ήθελα να τονίσω από πλευρά των Πρασίνων. Είναι σημαντικό να ε, εντατικοποιηθούν οι σχέσεις με το Ιράν. Μιλάμε για μια στρατηγική σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ιράν. Θέτουμε και το θέμα της ε, επίτευξης, τελικής επιτευξής των, της συμφωνίας, ε, ελπίζουμε τουλάχιστον. Πολλές αποστολές εμπορικές ήδη έχουν λάβει χώρα, πολλές πολιτισμικές ανταλλαγές για να κατανοήσουμε καλύτερα οι δε και για να αποκτήσουμε μια καλύτερη αίσθηση του τι αισθάνεται ο πολίτης, ο απλός πολίτης για τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να ανοίξει την προσωπία στο και αυτό θα πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν ζήτησε από τον πρόεδρο τη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων να αποσταλεί μια, επίστολη όπου θα αναφέρεται ότι θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να ανοίξει αυτή η αποστολή και θα πρέπει να διατεθούν και τα ανάλογα κονδύλια. Δεύτερο σημείο που ήθελα να τονίσω, παρά το γεγονός ότι η έκθεση δεν ε, περιλαμβάνει λεπτομερή απαρίθμηση των θεμάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεμονωμένη αναφορά παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό είναι καλό. Θα πρέπει να ξεκινήσει παρόλα αυτά μια γενικότερη συζήτηση. Και θα πρέπει να γίνουν κάποια βήματα ως προϋπόθεση για μια τέτοια συζήτηση. Άρα υποστηρίζουμε το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με το Ιράν και διαφόρων ειδών ανταλλαγές και θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ανοίξει αυτή η αντιπροσωπεία. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο, να δώσω το λόγο στην κύριο Σαλαφράγκα, εφόσον το επιθυμεί. Ευχαριστώ. Θα ήθελα απλώ να πω ότι ω και όδηση γιατί τη ομάδα μου είχε σημαντικέ ε, υποχρεώσει στα πλαίσια των εκλογών. Θα ήθελα απλώ εκ μέρου του να πω ότι οι τροπολογίε του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ε, είναι ελαστικές, δείχνουν το συνεργάσιμο πνεύμα μας φυσικά με σεβασμό των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και θα θέλαμε να εκφράσουμε τη συμφωνία μας με τις περισσότερες τροπολογίες της ομάδας και της ομάδας των μεταρρυθμιστών και συντηρητικών. Μια και απουσιάζει η συγγήτρια, δεν έχει νόημα να σας αναλύσω πιο διεξοδικά τη θέση του και όδους ως προς τις τροπολογίες. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να κάνω μια ενδελεχή ανάλυση της θέσης του Ισκιώδου Συγγετού για τις τροπολογίες ε, εν τη απουσία της εισηγητρίας. Ευχαριστώ κυρία Σάκη. Ευχαριστώ πολύ. Να τονίσω ότι Είμαι απογοητευμένη με το πώ εξελίχθηκαν τα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι όντω πρέπει να ψηφίσουμε αύριο, γιατί πρέπει να γίνει αυτό και να προλάβουμε εντό τη θητεία. Θα συμφωνήσω λοιπόν εδώ με τη σύστασή σα. Όμω, για την δική μου τροπολογία προς τη σύσταση προς το Συμβούλιο για μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις σχέσεις μας με το Ιράν ή τέλο παντών ως προς το Ιράν με την αντιπροσωπεία μας για το Ιράν τον περασμένο Δεκέμβριο και την επίσκεψη που κάναμε είδαμε τι δυνατότητες ανοίγματο υπάρχουν εφόσον πάρουν σαρκοκευστά πέραν των τεχνικών διαπραγματεύσεων περί των πυρηνικών κάτι στο οποίο κανένα από τα μέλη μας δεν συμμετέχει επί της ουσίας, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν μια από τις πρώτες μας προτεραιότητες και μου ξεκινούν από την έμφαση στην τόνωση της ελευθερίας των γυναικών ως προς την ελευθεροτυπία, την ελευθερία της έκφρασης και το ρόλο του δικαστικού κλάδου. Το γεγονός ότι πολύ συχνά οι υποπτοί δεν έχουν δυνατότητα νομικής αρρωγής και οι δίκες ε, ολοκληρώνονται πολύ γρήγορα με σοβαρότατες καταδίκες όπως ε, ε, πολλές φορές η εκτέλεση διαδικασίε. διαδικασίες. Ε, Επίση, ελέγξαμε και την κατάσταση στο Αφγανιστάν και το τι έγινε μετά το τέλο τη χρονιά Η ροή εμπορίων ναρκωτικών και τα παράνομα, η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών μέσω του Ιράν προ περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που μας απασχόλησε. Είδαμε κατά πόσο μπορεί να υπάρξει δυνατότητα να διερευνήσουμε τρόπου συνεργασία. Αλλά με τη σαφή προπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν συλλήψεις υπόπτων με ευρωπαϊκή ανάμειξη που να οδηγήσουν ενδεχομένως και σε θανατώσεις. Εφόσον συνεργαστούμε με τις Ιρανικές αρχές δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να υπάρχει τέτοιου είδους τιμωρία. Από την άλλη υπάρχει και κοινή ευθύνη για το τι θα γίνει μετά την αποχώρηση των ε, δυνάμεων της Δύσης από το Αφγανιστάν. Ξέρουμε ότι στο Ιράν υπάρχουν και εκατομμύρια Αφγανοί πρόσφυγες σε μια χώρα που είναι ήδη ευάλωτη. Πολλά από τα ζητήματα όπως οι ανταλλαγές φοιτητών και άλλα ζητήματα που απασχολούν τους μεν και τους δε είναι κάτι που καλύτερα θα τα κάλυπτε μια ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία, αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτόπου. Όντως, τέτοιες εντονισμένες προσπάθειες θα έχουν διαρκή αποτελέσματα και πιο θετικά σε σχέση με τις μεμονωμένες προσπάθειες όπως αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε την δυνατότητα ανοίγματο όπως ε, φάνηκε μέσα από τις πρώτες της εκφράσεις στο ζήτημα των πυρηνικών, αλλά θα πρέπει να μην φανούμε και αφελείς, διότι υπάρχουν ζητήματα που όντως είναι πολύ ε, δυσχεροί, αποτελούν πρόσκομα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από την πλευρά των Ιρανικών αρχών. Είναι η κατάσταση στη Ρωσία, στην, η, ο πόλεμος στη Συρία θα πρέπει να δοθεί ένα τέρμα εδώ, να δοθεί τέρμα στον τρομακτικό πόνο των ανθρώπων, εκατομμύρια γυναίκες και παιδιά που είναι τόσο ευάλωτοι. Εδώ στη Συρία το Ιράν διδραματίζει έναν πολύ επιζήμιο ρόλο με τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χεσμολάχ που ε, δεν επιτρέπουν την πάυση των εχθροπραξιών. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί ένα τέρμα στις τρομοκρατικές ενέργειες στην περιοχή και να ε, δούμε και το θέμα των μαζικής καταστροφής από αυτή τη σκοπιά. Μπορεί να περιληφθεί στις ατζέντε των συνομιλιών μας με τους Ιρανούς και στο μέλλον. Αυτές είναι λίγο πολύ οι τροπολογίες που υποβλήθηκαν και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα κοινό ψήφισμα με ηχηρές δηλώσεις για το μέλλον της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράν. Για το ποιο θα πρέπει να είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα ε, και να είμαστε ρεαλιστές αλλά και πραγματιστές. Δηλαδή να προωθήσουμε τα ευρωπαϊκά ζητήματα αλλά να επιδιώξουμε και βήματα προόδου και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον πόλεμο στη Συρία και την διακίνηση ναρκωτικών αλλά και την κατάσταση των προσφύγων. Εκεί πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε και νομίζω ότι θα έχουμε αύριο μια επικοδομητική ψηφοφορία πληροφορία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Ο κύριο Τάνοκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα η ομάδα μου είναι αρκετά επιφυλακτική και λιγότερο πιεστική στις σχέσεις με το Ιράν. Ο κύριος Ροχάνη έδειξε μια αλλαγή στη στάση του και έχει φανεί ένας αγγελιοφόρος καλών ειδήσεων. Νομίζω λοιπόν ότι καλόπιστα έχουμε διαπραγματευτεί ω τώρα μαζί του και βεβαίω υπάρχει και ένα ρεύμα σκέψη που λέει ότι όλα αυτά μπορούν να είναι περαστικά. Η νέα λοιπόν συμφωνία είναι καλή ε, εφόσον όμω οδηγήσει σε πραγματική πάυση του πυρηνικού προγράμματο. Προ στιγμήν αυτό δεν φαίνεται να είναι κάτι που θα συμβεί άμεσα. Ε, Επίση, έχουμε κάποιε επιφυλάξει για το κατά πόσον μπορεί το Ιράν να συμμετάσχει ω ένα ε, ισότιμο εταίρο στι ε, συνομιλίε για την εξέλιξη για το μέλλον στη Συρία. Δεν θέλουμε να δοθεί υπερβολικά μεγάλο βάρος στο ρόλο του στην πάυση του εμφυλίου αυτού πολέμου. Και επίσης για την αντιπροσωπεία στο Ιράν. Ίσως είναι διαφορετικό αυτό από το να υπάρχει απλώς ένας σταθμός ή μια υπηρεσία της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Όλα το να υπάρχει συγκεκριμένο γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεία ίσως είναι σαν να λέμε στο Ιράν ότι τους αποδεχόμαστε. Τους αποδεχόμαστε παρά τις αποτρόπες ε, ε, τα του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, με την δίωξη ανθρώπων για τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις, τις τιμωρίες σε ανηλίκους, την δίωξη των θρησκευτικών πεπιθήσεων και ούτω καθεξής. Ευχαριστούμε κύριε Σκουάντρας. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η προφύλαξη θα πρέπει να είναι η κατευθυντήρια γραμμή μας ε, και η επιφυλακτικότητα σε ό,τι αφορά τις συστάσεις μας για το Ιράν. Έχουμε τη συμφωνία του Νοεμβρίου της Γενέβης, του Νοεμβρίου του 2013, πολύ σημαντική συμφωνία. Αλλά όπως δείχνουν και οι τροπολογίες που έχω προσυπογράψει μαζί με τον Τούνα Κέλαμ και άλλα μέλη της ομάδας, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι το Ιράν εξακολουθεί να παραβιάζει πολλά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συνθήκη για τη μη διάδοση των όπλων. Δεν θα πρέπει να σπεύσουμε λοιπόν να άρουμε τις, ε, τους περιορισμούς. Απλώς ε, ευελπιστούμε ότι αυτή η ενδιάμεση συμφωνία θα μας οδηγήσει σε μια τελική, οριστική, περιεκτική και σφαιρική συμφωνία. το Ιράν με την αποφυλάκηση κάποιων πολιτικών κρατουμένων ή κρατουμένων για λόγους συνείδησης τον περασμένο Σεπτέμβριο έκανε μια θετική χειρονομία. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να μας κάνει να θελοτυφλούμε μπροστά σε πολλές άδικες δίκες, εκτελέσεις, αδικαιολόγητες συλλήψεις, καθώς και βασανιστήρια πολιτικών ακτιβιστών ή μελών μειονοτήτων. Γιατί αυξήθηκαν δραματικά οι εκτελέσεις μετά την ανάληψη του υποτιθέμενου μετριοπαθούς Ρουχάνη. Και μάλιστα τις πρώτες δύο εβδομάδες του έτους 40 άνθρωποι απαχωνίστηκαν. Δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε λοιπόν αυτή τη σημαντική αύξηση των εκτελέσεων. Επίσης θα πρέπει το Ιράν να δώσει χορήγηση διαβατηρίου στον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών για το Ιράν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί είχα συνάντηση με την κυρία Σιρήνε Μπαντή, βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Τη συνάντησα στο γραφείο μου και μου επισήμανε τη σπουδαιότητα που έχει αυτό το σημείο. Δηλαδή, αν ο ειδικό απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ε, μπορέσει να μεταβεί στο Ιράν, δεν επιτρεπεί επιτρεπεί είσοδο στο Ιράν για να εργαστεί επιτόπου, τότε γιατί μιλάμε. Η συμβαστική τροπολογία αναφέρει ότι θα πρέπει να στηρίξουμε το έργο του ειδικού εισηγητού των Ηνωμένων Εθνών για το Ιράν αυτή η διατύπωση όμως παρά είναι αόριστη. Θα πρέπει να απαιτήσουμε από το Ιρανικό καθεστώς να χορηγήσει στον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα θεώρηση διαβατήριου για να μπορέσει ο ειδικό εισηγητή να μεταβεί στο Ιράν και να κάνει έρευνα επιτόπου για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν δεν απαιτήσουμε κάτι τέτοιο, κάνουμε μια τρύπα μέσα στο νερό. Τέλο, η σύσταση, η πρόταση να συμμετέχει και το Ιράν στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων για την επίλυση της ε, κρίσης στη Συρία ε, δείχνει ότι αγνοούμε ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να είναι τμήμα της λύσης. Γιατί το Ιράν εξακολουθεί να στηρίζει ενεργά το καθεστώς του Ασάτ. Πώς το καλούμε λοιπόν στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Οπότε θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν απερίσκεπτο. Έχουμε μια ενδιάμεση συμφωνία Ας περιμένουμε λοιπόν για να διαπιστώσουμε το κατά πόσο το ΙΡΑ θα εφαρμόσει αυτές τις διατάξεις και πραγματικά θα κάνει βήματα προς περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη συνεργασία. Ευχαριστώ ο Σερ Ρόμπερτ. Α, δεν ζήτησε το λόγο. Δεν ζήτησε το λόγο. Ήταν ε, ανακριβής οι μου λοιπόν. Θα ήθελα και εγώ να σας μεταφέρω κάποια σχόλια που μου διαβίβασε στο μεταξύ η Μαρία. Θα στα διαβάσω μάλιστα. Έχουμε εδώ τρία βασικά σχόλια, τρία βασικά σημεία. Ξέρετε ότι η ομάδα θα, μας, θα καταψηφίσει την τροπολογία 73 που διαγράφει το, την έκκληση για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας στο Ιράν. Υπάρχει διάσταση απόψεων εδώ μεταξύ των πολιτικών ομάδων, το γνωρίζουμε. Άκουσα τις απόψεις, θα τις διαβιβάσω στην εισηγήτριά μας, την κυρία Μαρία Μουνής. Επίσης, η τροπολογία 156 που ε, εξαρτά τις διακοινοβουλευτικές μας ε, συναντήσεις στο Ιράν από συναντήσεις με τις εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών παρόλο που συμφωνούμε ότι η αντιπροσωπεία θα πρέπει να έχει συναντήσεις με την ε, ε, κοινωνία των πολιτών, το να θεωρούμε αυτή την επαφή ως εκ των όνων προϋπόθεση και να εξαρτούμε από αυτό την σύσταση της, ε, την πραγματοποίηση της αποστολής, θεωρούμε υπερβολικό. Επίσης, ε, η αναφορά των ψηφισμάτων του ΟΗΕ δεν είναι χρήσιμη γιατί τα ίδια τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας έχουν αυτή τη στιγμή διαπραγμάτευση με το Ιράν και αποκλείουν ουσιαστικά από τα προηγούμενα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Οπότε έχουμε κάποια διαφορά μεταξύ των έργων και των λόγων. Αυτά τα τρία σημεία μου επισημαίνει η, η συγγήτρια ως ε, σημαντικά. Αύριο θα έχουμε τη σχετική ψηφοφορία και θα λυθεί η απόφαση σχετικά με τη σύσταση. Περνάμε τώρα στην επόμενη έκθεση της κυρίας Όγιλον που επίσης απουσιάζει αλλά ο Σερ Graham Βότσον θα την αντικαταστήσει και θα μας παρουσιάσει τη σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την καθιέρωση κοινών περιορισμών όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων στους αξιωματούχους της Ρωσίας που ενέχονται στην υπόθεση Σεργέη Μαγνίτσκι. Τώρα θα έχουμε σε λίγο πρόβλημα για ποιου λόγου ε, αρνούμαστε τη χορήγηση θεώρηση διαβατηρίων ε, σε ε, Ρώσοι εξαιτία κρυμαία, εξαιτία υπόθεση υπόθεσης Μαγνίτσκι. Θα πρέπει να βρούμε και την νομική βάση. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η συνάδελφο, η κυρία Όγιουλαν, λυπάται που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Όμως, είχε επαφέ με του την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο και νομίζω ότι έχουμε εδώ μία σύσταση η οποία μπορεί να ψηφιστεί αύριο ε, κιόλα. Νομίζω ότι υπάρχει γενικώ στήριξη για να έχουμε και ένα κατάλογο με ονόματα, αλλά ίσως να μην έχουμε τη στήριξη των σοσιαλιστών και δημοκρατών ακριβώς για το σημείο αυτό. Νομίζω το μόνο μέλος της ομάδας αυτής που είναι και ε, μην τον κολακεύετε, ε, το μόνο... Μην πυροβολείτε τον πιανίστα. Νομίζω όμως ότι ο κύριος ε, Βράντα ήταν ένας από τους πελάτες του κύριου Μαγνίτσκι υπό κάποια έννοια, διότι πραγματικά έφερε, ε, διοργάνωσε μια ολόκληρη εκστρατεία για τον κύριο Μαγνίτσκι για τα μέλη της οικογένειάς του, ώστε να δικαιωθεί. Πάντως, Πρόεδρε, θα γνωρίζετε ότι την ε, σύσταση αυτή ε, την πρότεινα ήδη από το Φεβρουάριο του 2012 στην Επιτροπή αυτή, ώστε να υπάρχει μια συνεκτική πολιτική έναντι καθεστώτων κατά των οποίων λαμβάνουμε μέτρα ε, αντιπίνων. Έτσι, από τον Οκτώβριο του 2012 γίναμε μια πρώτη σύσταση για την ε, πρόβλεψη κοινών περιορισμών στην έκδοση θεωρήσεων για Ρώσους αξιωματούχους που ενέχονταν στην υπόθεση Σεργέ Μαγνίτσκι. Αυτό συνέπεσε με μια παρόμοια πρωτοβουλία από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών να προβλέψουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς έναντι των ίδιων αξιωματούχων και άλλων προσώπων που ενέχονταν σε περιπτώσεις παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία. Στη σύστασή μα, από τον Οκτώβριο του 2012 καλούσαμε το Συμβούλιο να καταρτήσει ένα κατάλογο ακριβώ αυτών των Ρώσων αξιωματούχων που ενέχονταν στην ε, περίπτωση του ε, Σεργέη Μαγνίτσι και να του προσθέσει σε, μια, ε, σε ένα κατάλογο, σε μια λίστα απαγόρευση έκδοση θεωρήσεων. Όμω δεν αντέδρασε το Συμβούλιο, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εξωτερική δράση, ούτε είπατε εκπρόσωπο, το αίτημα αυτό και δεν έθεσαν στον κατάλογο προτεραιοτήτων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων το όλο θέμα. Ούτε ενημέρωσαν το Κοινοβούλιο για τις δράσεις που ανέλαβαν. Αυτό είναι κάτι το οποίο με τη στήριξή μα έφερε λοιπόν παρά στην προσοχή της, ε, έφερε πάλι στην προσοχή της Επιτροπής μας η κυρία Όγιουλαντ και Ακριβώ γι' αυτό κλείθηκε η Ολομερία να ψηφίσει για το κείμενο τη σύσταση. Υπάρχουν 32 ονόματα στην ε, σύσταση αυτή και η συμβαστική λύση με τον εισηγητή του ΕΛΚ ώστε στην παράγραφο 1 αντί να προσθεθεί εξή διατύπωση και νομίζω το κείμενο έχει μοιραστεί στου συναδέλφου. Λέει ότι βάσει τη λογοδοσία ε, και του νόμου για λογοδοσία στα πλαίσια του 100 από το 2012 θα πρέπει μεταξύ άλλων να προστεθεί στον κατάλογο απαγόρευση έκδοση θεωρήσεων για Ρώσους, για πολίτες να προστεθούν τα εξή ονόματα. Η συμφωνία αυτή αφήνει περιθώριο στο Συμβούλιο για περαιτέρω προσαρμογές και προσθήκες στον κατάλογο Πάντως, στον κατάλογο αυτό προβλέπονται τα 16 πρόσωπα, τα οποία περιλαμβάνονται και στον κατάλογο απαγόρευσης από τις ΗΠΑ καθώς και 16 ακόμη άνθρωποι, οι οποίοι συμμετείχαν στις ε, μεταθανάτιες ε, δίκες κατά του κυρίου Μαγνίτσικη και των μελών της οικογένειάς του. Από πολιτική σκοπιά τώρα, βεβαίω αναγνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη, περισσότερο από ότι το Ευρωκοινοβούλιο, είναι αρμόδιοι, είναι το σώμα, το σώμα που πρέπει να αποφασίσει για την. Ε, το θεσμικό όργανο πρέπει να αποφασίσει για την απαγόρευση έκδοση θεωρήσεων, όπω και για την αναθεώρηση των συνθήκων. Πιστεύω όμω ότι πρέπει να αντιδράσουν βάσει των συστάσεων που έχουμε εγκρίνει στον, ε, στο θέμα αυτό. Η σύσταση αυτή έχει περισσότερο συμβολική αξία, αλλά έχει τη σημασία τη είναι η στιγμή να δείξουμε ότι οι εγκληματίες και οι παραβάτες δεν μπορούν να υποφελούνται των ταξιδιωτικών διευκολύνσεων, της πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές και άλλες υπηρεσίες, όπως τους αρέσει, ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγκρίνοντας τη σύσταση αυτή, στέλνουμε δύο σοβαρά πολιτικά μηνύματα. Ένα προς το Συμβούλιο, ώστε να λαμβάνουν υπόψη του σοβαρότατα τέτοιου είδου συστάσει το ίδιο και την είπατε εκπρόσωπο, και κατά δεύτερον ε, στου πολίτε τη Ρωσική ε, Ομοσπονδία. Ότι μπορούμε να επιδείξουμε αλληλεγγύη, αλλά και πυγμή στον, στην αντίθεσή μα κατά των ενεργειών της ομάδας εγκληματιών, της συμμορίας που καμιά φορά ε, μπορούμε να πούμε ότι έχει τα ενία της διακυβέρνησης στο Κρεμλίνο. Πρόεδρος. ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον αναπληρωτή της κυρία Σόγιουλα, τον κύριο Γουάτσον, που μας έκανε την παρουσίαση της ε, σύστασης της έκθεσης. Εκ μέρους του ΕΛΚ θα ήθελα να πω ότι εμείς ε, ταχθήκαμε υπέρ της συμπερίληψης του θέματος αυτού στην ημερήσια διάταξη, γιατί πιστεύουμε ότι ρητά θα πρέπει και κατηγορηματικά να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι σε τέτοιες ε, καταστάσεις. Και Εδώ προτείνεται ε, η συμπερίληψη του συγκεκριμένου καταλόγου και ο κύριος Πρωτασέβης, ο σκιώδης ηγητής μας, ε, συμφώνησε με την εισηγητή ότι συμφωνούμε να συμπεριληφθεί ο κατάλογος με τα 32 ε, πρόσωπα με την προσθήκη μεταξύ άλλων, ώστε να εξεταστεί και από το Συμβούλιο η πρόταση αυτή έχουμε αποσύρει τις σχετικές τροπολογίες και αύριο θα υπερψηφίσουμε την έκθεση κυρία Σόγιουλαντ ε, που έχει το περιεχόμενο που μας περιέγραψε ο κύριος Γουάτσαν. Ευχαριστώ κυρία Λόχπιλερ. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι εξ ονόματο των Πρασίνων υποστηρίζουμε και εμεί τη σύσταση και ίσω θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η σημερινή απόφαση επί των κυρώσεων. Γιατί ένα τμήμα των κυρώσεων για την Κρυμαία αφορά ακριβώς τα ίδια θέματα και τις ίδιες κυρώσεις που ζητούμε και στην ε, υπόθεση Μαγνίσκη. Αυτό θα το ανακαλύψουμε όμως στην, ε, με την πάροδο της εβδομάδας. Κύριε Γκράμα, θέλετε να πάρετε, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φυσικά ξέρουμε ότι το Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να επιβάλλει περιορισμούς σε ό,τι αφορά τα ταξίδια και πάγωμα ε, κεφαλαίων σε ό,τι αφορά πράξεις που απειλούν την εδαφική αικαιρεότητα ή την κυριαρχία της Ουκρανίας. Ε, αναρωτιέμαι κατά πόσον ε, οποιαδήποτε από τα άτομα είναι τα ίδια άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση Μαγνίτσκι. Η παρατηρήση που κάνετε εξ αρχής, ε, πρόεδρε, στην αρχή της συζήτησης ιδια ατομα που εμπλέκονται στην υποθεση μαγνιτσκι η παρατηρηση που πραγματικά μια πάρα πολύ επίκαιρη παρατηρήση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ψηφίζουμε λοιπόν αύριο. Και τώρα να περάσουμε στο τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η έκθεση Κρίστοφ Λίσεκ για τη συμφωνία πλαίσια μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας. Και επειδή δεν υπάρχουν ουσιαστικά τροπολογίες εδώ, νομίζω ότι ξέρετε ότι στο σημείο αυτό δεν υπάρχει ανάγκη για συζήτηση. Αύριο θα γίνει η ψηφοφορία για το θέμα αυτό. Οι συζητήσει, η ψηφοφορία θα ξεκινήσει αύριο 9 και 4. 9 και 4. Σε Ρόμπερτ. Τι σημαίνει αυτό, ότι στι 9 όλοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν. Μάλιστα λοιπόν, ολοκληρώθηκε έτσι η συνεδρία. Τα λέμε λοιπόν αύριο κυρίε και κύριοι. Σα ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.